Καλημέρα σας όλες σας. Αρχίζουμε. Με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχει μια αλλαγή στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης στο σημείο 15, δηλαδή η συζήτηση για την γνωμοδότηση του κυρίου Μπούγκα πολέμηση της παράνομης αλληλείας σε παγκόσμιο επίπεδο θα εξεταστεί σήμερα αντί για το σημείο 4. Το δε σημείο 4 έκθεση του κυρίου Κασμάρεκ αύξηση της επίπτωσης της πολιτικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναβληθεί για αύριο το απόγευμα μετά τις ψηφοφορίες. Το δε σημείο 11 αναβάλλεται για αύριο το τέλος της πρωινής συνεδρίας έτσι ώστε ο κύριος Σικλούνα να μπορέσει να προσέλθει. Μήπως υπάρχει καμία αντίρρηση στις αλλαγές αυτές της ημέρησης διάταξης. Όχι, ε, τότε εγκρίνεται. Δύο ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Λάβαμε ερωτήματα της κυρίας Σαργεντίνη για την πράσινη βίβλο της Επιτροπής επί της Μελλοντικής Πολιτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ερωτήσεις αυτές έχουν διανεμηθεί γαλλικά και αγγλικά. Δώνω λοιπόν το λόγο στην Κομισιόν για να απαντήσει στις ερωτήσεις της κυρίας Σαργεντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Ολίβιος Μοδέρν. Από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας. Τα ερωτήματα της κυρίας Αργεντίνη αφορούσαν τα δύο πρώτα τους λόγους και τους σκοπούς της διαδικασίας που άρχισε μετά την έγκριση της Πρασίνης Βίβλου από την Κομισιόν στα τέλη του χρόνου και που κατέληξε στην έγκριση σε εφέτος για το μέλλον της αναπτυξιακής παλιτικής. Το θέμα αυτό βασικά λοιπόν είναι αν η αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης μπορεί και πρέπει να ενημερωθεί για να ληφθούν υπόψη οι σημερινές προκλήσεις και να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα του φορολογουμένου και της φορολογουμένης θα χρησιμοποιούνται όσο δυνατόν αποτελεσματικότερα με βάση τους στόχους της συνεργασίας. Για τη διαβούλευση ως προς την πράσινη βίντεο έγιναν διαβουλεύσεις μετά τη δημοσίευσή της η τελευταία έληξε τον Ιανουάριο του 2011 και κατέληξε σε πολλές συνεισφορές από μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων και αυτά όλα θα τροφοδοτήσουν την ανακοίνωσή μας του Μαΐου η οποία θα καθορίζει τα πλαίσια της μελλοντικής πολιτικής ανάπτυξης και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή των επομένων δημοσιονομικών προοπτικών μεσοπρόθεσμα. Τώρα, για ποιους λόγους οθήθηκε η Επιτροπή να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. Η συγκυρία άλλαξε ως προς την ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στην Ένωση. Εμφανίστηκαν νέοι δωρητές, ε, καινούργιες προκλήσεις όπως οι κλιματολογικές αλλαγές μαζί με την πρόκληση της τροφιμικής ασφαλείας και συνέχιση η παράταση της ανέχειας. Η πίεση επί των δημοσιονομικών των χωρών μελών δεν επιτρέπει να λύσουν αυτά τέτοια προβλήματα. Και η εξωτερική και εσωτερική τέτοια πίεση καθιστά απαραίτητη την εκμετάλλευση όλων των δυνατών δρόμων ώστε η αναπτυξιακή πολιτική να έχει όσο δυνατόν με καλύτερες, περισσότερες επιπτώσεις ως προς την καταπολέμηση της ανέχειας. Το τρίτο <coughs> ερώτημα της κυρίας Αργεντίνη αφορούσε τον ορισμό που θα ήταν μία συμπεριληπτική λέει ανάπτυξη που να συμπεριλαμβάνει δηλαδή και τους πτωχούς και τους ανέργους και με ποιο, ποια μέσα θα μπορούσε να εφαρμοστεί ή μάλλον τους ηλικιωμένους και τους πτωχούς. Για τη μείωση της ανέχειας Πράγματι θα έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια συμπερίληψη διότι θα επέτρεπε σε όλους να υποφεληθούν. Μια τέτοια συμπεριληπτική ανάπτυξη θα μπορούσε να δημιουργήσει και περισσότερες θέσεις εργασίας και άρα θα επέτρεπε με καλύτερη συμμετοχή του πληθυσμού στις δραστηριότητες έρευνας αλλά και στην καταπολέμηση της ανέχειας η μελλοντική αναπτυξιακή μας πολιτική θα συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Το τέταρτο ερώτημα αφορούσε τα μαθήματα που πήρε η Κομισιόν από το παρελθόν και ως προς την πολιτική συνεργασία της και ως προς τη συνοχή των αναπτυξιακών της προγραμμάτων. Για το πρώτο από αυτά τα δύο τελεταρτα ερωτήματα θα ήθελα να πω ότι εφαρμόζουμε τις αρχές της δήλωσης της Άκρας και των Παρισίων ιδιαίτερα δε ιδιαίτερα δε μία από αυτές. Όλα αυτά γίνονται σε σενή συνεργασία με τις αρχές των διαφορεμένων χωρών που ευθυγραμμίζονται με τα αναπτυξιακά του σχέδια. Τελεία. Όσο για τη συνοχή των αναπτυξιακών προγραμμάτων στις ε, αναδυόμενες χώρες, εμείς ε, προωθούμε οποιοδήποτε τέτοιο σχετικό διεθνές πρόγραμμα, γιατί η αρχή της συνοχής των αναπτυξιακών προγραμμάτων έχει επαναληφθεί πολλές φορές και το 2005 στη συνθήκη της Λισαβόνας ιδιαίτερα. Τη θεωρούμε προτεραιότητα. Όπως τις διαδικασίες, η Επιτροπή καθορίζει κανόνες εσωτερικής της λειτουργίας, αξιολογήσεις και πρόγραμμα εργασίας που βασίζεται στο δικό της εσωτερικό πρόγραμμα έτσι ώστε να ταυτιστούν καλύτερα οι στόχοι και οι δραστηριότητες που έχουν μεγαλύτερη συνέπεια με την εγκεκριμένη αναπτυξιακή πολιτική. Οι πρόοδοι που θα έχουν σημειωθεί στην Ένωση αξιολογούνται από την Κομισιόν και αποτελούν ακόμη ένα εργαλείο εφαρμογής της συνοχής. Η επόμενη τέτοια έκθεση θα υποβληθεί τον Οκτώβριο του 2011 και θα είναι η τρίτη τη αυτή. Το Κοινοβούλιο, εάν θέλει, μπορεί και αυτό να συμβάλλει στην έκθεση αυτή. Τώρα ως προς την ουσία. Πολλά παραδείγματα δείχνουν ότι έχουν σημειωθεί πρόοδοι ως προς τη συνοχή αν και μπορούν ακόμη να γίνουν βελτιώσεις και χρειάζονται περισσότερες διευθετήσεις. Έτσι παραδείγματο χάρη η πρωτοβουλία για την εφαρμογή των δασοκομικών κανονισμών για τις εμπορικές συναλλαγές που λέγεται FLECT σκοπεύει να συνδυάσει την κλιματολογική πολιτική με την αναπτυξιακή. Για τα τρόφιμα έχουμε πει ότι οι επιχορηγήσεις που δίνονται από την ΚΑΠ και η κατάργηση, σχεδόν κατάργηση των επιστροφών προς τις εξαγωγές έχει διορθώσει τις τρευλώσεις του παρελθόντος. Για την αναθεώρηση της ΚΑΠ και της αλληλείας, της πολιτικής της αλληλείας, Ξανασκεφτήκαμε τους αναπτυξικού μας στόχους ιδιαίτερα ως προς την τροφιμική ασφάλεια. Και τέλος η Κομισιόν τελευταία ενέκρινε δύο ανακοινώσει δύο ανακοινώσει, τη μία για την πρόσβαση στις πρώτε ύλε που συμπεριλαμβάνει και ένα μεγάλο τμήμα για την ανάπτυξη και την άλλη ως προς τη φορολογία. και ακόμα επεξεργαζόμαστε τα μέσα με τα οποία θα μπορούσαμε να ταυτίσουμε τους καλύτερους τρόπους για να βελτιστοποιηθεί η φορολογία και η ανάλυση αυτή γίνεται χώρα με τη χώρα και δεν αγνοεί και την ε, διαφάνεια που πρέπει να υπάρχει στις επιχειρησιακές δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μήπως η Κομισιόν θέλει να μας δηλώσει τίποτα ως Επιτροπή Αναπτύξεως. Όχι. Α, καλά τότε. Σημείο 5. Χρηματοδότηση της Ένωσης για το μέλλον. Εδώ προβλέπεται ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Γιούτα Χάουγκ πρόεδρο της Επιτροπής ΣΥΡ. Τον Ιούνιο η Επιτροπή αυτή, η ειδική δηλαδή Επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τις δημοσιονομικούς πόρους της Ένωσης μετά το 2013 θα αποφανθεί για το δημοσιονομικό πλαίσιο 14-20. Η έκθεσή της λέγεται «Επενδύσεις στο μέλλον δύο ένα νέο πλαίσιο πολιετές πλαίσιο χρηματοδότησης για μια Ευρώπη ανταγωνιστική, βιώσιμη και συμπεριληπτική. Εμείς έχουμε εγκρίνει ήδη μία έκθεση, την έκθεση της Μπέρμαν, έτσι ώστε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας μέσα στα πλαίσια το στόχο της χιλιετίας για την ανάπτυξη και για να αναπτύξουμε το κεφάλαιο εξωτερική πολιτική που προσδίδει μεγαλύτερη ευελιξία και νέες πρωτοβουλίες σε σχέση με την ανάπτυξη ενός, ενός νέου πλαισίου χρηματοδότησης, ιδιαίτερα ενός φόρου για, τους, για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους πλέον πτωχούς και να εγγυηθούμε την συνοχή των ε, πολιτικών ανάπτυξης. Είχαμε ήδη μία ανταλλαγή απόψεων με τον ε, εισηγητή της ΣΥΡ, τον κύριο Γκαρίγκα, όμως τον προηγούμενο μήνα οι συντονιστές αποφάσισαν να γίνει μια νέα συζήτηση επί του θέματος με την κυρία Γιούτο ε, Χάουγκ, πρόεδρο της ΣΥΡ. Την καλωσορίζω και θα θέλαμε να μας πείτε πώς εσείς και οι συνάδελφοί σας ε, συμμερίζεστε τις ιδέες μας και τη γνωμοδότησή μας. Κυρία Χάουγκ, έχετε το λόγο. Ähm, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία για την πρόσκληση. Από την αρχή εγώ έλεγα ότι η ενημέρωση είναι ε, σημαντική για όλες τις επιτροπές διότι αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει μια γνωμοδότηση θα πρέπει να αποφεύγουμε να προορίζεται αυτό στους 52 βουλευτές της Επιτροπής της συγκεκριμένη, αλλά όλοι οι συνάδελφοι να είναι έτοιμοι για τον Ιούνιο στην Ολομέλεια να μπορέσουν από κοινού να εγκρίνουν τη θέση του Κοινοβουλίου. Διότι μόνο άμα κάνουμε κάτι από κοινού με μια μεγάλη πλειοψηφία μόνο έτσι θα μπορούμε να έχουμε το ειδικό βάρος για να περάσουμε την θέση μας στο Συμβούλιο. Τα πράγματα όμως δεν είναι και τόσο εύκολα. Έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης μπροστά μας. Η συνάδελφός μας έκανε μια, ένα σχέδιο ε, εκθέσεως που έχει 122 παραγράφους. Επαναλαμβάνω 122. Και αυτό το σχέδιο εκθέσης δεν ξέρω ποιος είχε τη δυνατότητα ήδη ε, ή το ενδιαφέρον να το δει, αλλά στηρίζεται σε έξι τομείς, σε έξι κεφάλαια. Το πρώτο έχει να κάνει με τις προκλήσεις. Το δεύτερο έχει να κάνει για μια καλύτερη εφαρμογή του κοινοτικού προπολογισμού και του ορισμού του προπολογισμού. Το τρίτο κεφάλαιο έχει να κάνει με τις προτεραιότητες, τις πολιτικές αυτές και θέματα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση, τη δομή και τη διάρκεια των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών, για μετά το 2015 μιλάμε, σε ένα πέμπτο κεφάλαιο προσπαθούμε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να έχουμε το θέμα της έκθεσης σε σχέση με την εκτέλεση του προπολογισμού από τη μια και την ε, έσοδα από την άλλη και τους ίδιους σπόρες, όπως ε, συνηθίζουμε να λέμε. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα σύστημα το οποίο παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο και εμείς ενδιαφερόμαστε για τον προγραμματισμό της δημοσιονομικής αυτής πτυχής. Και μετά έχουμε το επόμενο κεφάλαιο το οποίο αναπτύσσει την ιδέα ότι θα ήταν καλό να μιλήσουμε με το Συμβούλιο για θέματα διαδικαστικά. Κυρίως διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τον προπολογισμό που βοηθούν στη βελτίωση των ε, μελλοντικών προοπτικών όσον αφορά τα δημοσιονομικά. Η, τον Ιανουάριο Επιτροπή Ανάπτυξης μας ε, ενημέρωση. Εμείς λάβαμε υπόψη τις παραγράφους όχι ότι τις εντάξαμε ολοκληρωτικά, αλλά τις είδαμε ε, σαν μια βάση, σαν μια γνωμοδότηση πτυχή της Επιτροπής σας. 82, 83, 86 σαν παράγραφοι έχουν ληφθεί υπόψη από τον εισηγητή. Έχουν να κάνουν με τη μείωση της φτώχειας. Και επίσης στο θέμα που έχει να κάνει με τις αξίες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Εγώ θα έλεγα αυτό είναι η αρχή ε, όπως το βλέπει ο εισηγητής. Στη συνέχεια έχουμε τις τροπολογίες που έχουν καταταθεί και οι οποίες θα, αρχίζουν να, θα αρχίσει η εξέτασή τους. Έχουμε πάνω από χίλιες ε, τροπολογίες όπως καταλαβαίνετε. Θα μιλήσουμε, θα συζητήσουμε μαζί στις μελλοντικέ τρεις ενεδριάσεις για να προσπαθήσουμε να βρούμε συμβαστικές τροπολογίες ή δυνατόν και φυσικά να τις ξεδιαλέξουμε για να έχουμε μια σωστή κατάληξη. Επίσης ήθελα να πω η ομάδα μου έχει καταθέσει τέσσερις τροπολογίες οι οποίες στην κυριολεξία πλήρως ε, έχουν να κάνουν με είναι η παράγραφη 7, 8, 9 και 14 της Επιτροπής Ανάπτυξης και της... η ομάδα μου της υιοθετεί, θα λέγαμε. Επίσης υπάρχει το ενδιαφέρον ε, να δούμε πώς είναι οι άλλες πολιτικές ομάδες και αν έχουν τη διάθεση να ψηφίσουν αυτές εδώ τις τροπολογίες ή αυτά τα, κείμενα, αυτά τα σημεία του κειμένου. Ε, όχι με την ε, ιδιότητα της Προέδρου, δεν είναι μόνο η Επιτροπή Ανάπτυξης που έχει γνωμοδοτήσει. Θα πρέπει λοιπόν οι Επιτροπές να ε, δουν αυτή την εκθεσή και στο μέτρο του δυνατού ε, και αν το επιτρέπουν και άλλες πολιτικές ομάδες να κοιτάξουμε να εντάξουμε όσο δυνατόν περισσότερα μέρη στην εκθέση αυτή. Ε, η πρόεδρος μας ρώτησε για πώς έχει η πρόοδος. Την επόμενη πέμπτη θα γίνει μια πρώτη συζήτηση και θεωρώ ότι το προσθέτω αυτό, ότι καθένας όποιος θέλει να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση, αυτός αυτή είναι ευπρόσδεκτη. Είμαστε μια ανοιχτή επιτροπή, αλλά φυσικά όπως πάντα, καταρχήν θα ακούσουμε αυτούς που είναι αρμόδιοι τη ομάδα μας, και στη συνέχεια οι συνάδελφοι που ζητούν το λόγο, θα ζητήσουν το λόγο, συγγνώμη, θα μπορέσουν φυσικά να συμβάλλουν, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, τις ιδιαίτερες ιδέες τους. Εμείς θα ψηφίσουμε 25-26 Μαΐου θα ψηφίσουμε την έκθεση και ελπίζω τότε να έχουμε εντάξει σε αυτή την έκθεση όσο δυνατόν περισσότερες συμπληρωματικές ε, παραγράφους από τις άλλες ομάδες και ελπίζω η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών να μπορέσουν να ψηφίσουν αυτή την έκθεση στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέρμαν τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα αγγλικά. Γιατί το κείμενο που έχω μπροστά μου είναι στα αγγλικά. Χαίρομαι που επισκέπτεται η Γιούτα Χάουκ την Επιτροπή μας. Είναι μεγάλη τιμή για μας και χαίρομαι επειδή η Γιούτα μας ε, εξήγησε ότι οι σοσιαλιστές παίρνουν τέσσερις τροπολογίες από την έκθεση Ντέιβι και από την, από την Επιτροπή Ανάπτυξης δηλαδή και όπως εξελίσσονται οι συζητήσεις στην Επιτροπή ΣΥΡ, πιστεύω ότι θα οδηγηθούμε σε μία έκθεση που για τα επτά επόμενα χρόνια θα ζητάει τα ίδια με απειροελάχιστες αλλαγές. Δεν υπάρχουν οράματα για το τι χρειάζεται η Ευρώπη, τι χρειάζεται να χρηματοδοτήσει κατά τον 21ο αιώνα, ούτε βασικές επιλογές για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Μιλάμε για προστασία ε, ε, συμφερόντων που προϋπάρχουν. Είναι πολύ ανησυχητικό βεβαίως για τις αναπτυξιακές πολιτικές, διότι πολύ λίγες αλλαγές θα επέλθουν τη στιγμή που ε, υφιστάμεθα μεγάλη χρηματοοικονομική πίεση, πίεση για χαμηλότερο προϋπολογισμό, από πού θα προέλθουν τα χρήματα. Δυστυχώς θα πληγούν οι εξωτερικές μας πολιτικές, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να γίνονται περικοπές σαν προϋπολογισμό που δεν πλήττει άμεσα τους φορολογούμενους και τους ε, πολίτες γενικά που μας εκλέγουν. Φοβάμαι λοιπόν, εκφράζω τους φόβους μου για το μέλλον του προπολογισμού αναπτυξιακής βοήθειας, διότι η έκθεση Γκαρίγκα είναι ιδιαίτερα σύντομη όσον αφορά τις εξωτερικές πολιτικές και τα προγράμματα δράσης. Πολύ λίγες παράγραφοι, καμία ανάγκη μέτρων για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και τίποτα δεν αναφέρεται ως προς την αύξηση της ε, στήλης 4 γιατί θα πρέπει να καταπολεμηθεί η φτώχεια, ιδιαίτερα στην υποσαχάρια Αφρική. Ακούω λοιπόν από την Επιτροπή ότι εκφράζονται φόβοι για την φθήνουσα πορεία του προϋπολογισμού. Και δεν νομίζω θα δώσει και μεγάλη μάχη η Επιτροπή. Θα δούμε στις αρχές Μαΐου θα γίνει μια διάσκεψη του Διευθυντηρίου της Επιτροπής για το πολιετές ε, σχέδιο χρηματοδότησης. Επίσης, στην έκθεση Γκαρίγκα, και ελπίζω να αλλάξει αυτό, δεν γίνεται λόγος χρηματοδότησης ανθρωπιστικής βοήθειας από μία ανεξάρτητη γραμμή του προϋπολογισμού μέσα στα πλαίσια της ΕΙΕΔ και ως προς τις ε, πολιτικές μας επιλογές. Δεν είμαι σίγουρος για την έκβαση αυτών των συζητήσεων, αλλά η Ιούτα Χάουγ είναι πρόεδρος Επιτροπής ΣΟΥΡ και ξέρουμε ότι θα δώσει πολύ μεγάλο αγώνα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Γκέρενς έχει το λόγο. Ευχαριστώ να ευχαριστήσω την κυρία Χάου που ήρθε εδώ στην Επιτροπή μας. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να οργανώσει κανείς τη συνογή των, συνοχή των εργασιών μας. Έχω εκτιμήσει πάρα πολύ το ταλέντο της κυρίας Χάου και τον τρόπο με τον οποίο προεδρεύει. Κάποιες παρατηρήσεις. Είχαμε ευκαιρίες να μιλήσουμε μεταξύ μας, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε τη συζήτηση, επαναλαμβάνω, η πρώτη έχει να κάνει με την πολιτική συνεργασία και την ανάπτυξη. Αυτή η, πολιτική ε, πρέπει, είναι πανά να το πούμε, πρέπει να στοχεύει στην καταπολέμηση της στόχιας. Υπάρχουν παρά προβλήματα, κυ, κυρίως ότι έχουμε διασπορά των πιστώσεων, των πόρων, ε, και σε χώρες οι οποίες καταρχήν δεν έχουν επιλεχθεί στα πράγματα πρόγραμμα βοήθειας Σήμερα το πρωί συνάντησα εκπροσώπους της Concord και είδαμε τον τρόπο τον οποίο προσεγγίζουν το πρόβλημα. Τι κάνουνε. Επικεντρώνονται, το ενδιαφέρον σε προβλήματα σε χώρε όπου υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα φτώχεια ή σε χώρε οι οποίε έχουν γενικότερα πρόβλημα φτώχεια. Ε, και το θέμα είναι πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό. Πώς θα προχωρήσουμε. Θα κάνουμε μια παράλληλη προσπάθεια ε, τη στιγμή που δεν έχουμε πολλές φορές την ικανότητα να καταπολύσουμε τη φτώχεια σε συγκεκριμένες χώρες. Υπάρχουν επίσης χώρες οι οποίες έχουν μέσα, δημιουργούν πλούτο και μπορούν από μόνες τους, στα πλαίσια των συνόρων τους, να καταπολύσουν οι ίδιες χώρες τη φτώχεια όταν είναι σε ένα μέρος της χώρας. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε θέση πάνω σε αυτό. Είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε παλιότερα όσον αφορά το θέμα για τα μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη βοήθεια ανάπτυξης. Επίσης να πω και με την παρουσία εδώ της κυρίας Χάουγκ να πω ότι υπάρχει μια συνένεση όσον αφορά το πρόβλημα για τα χρήματα που επενδύονται σε σχέση με τις κλιματολογικές αλλαγές στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Πώς θα προχωρήσουμε. Θα προσθέσουμε και άλλους πόρους. Και πώς θα γίνει η χρήση αυτής της βοήθειας. Αυτό θα έχει σημασία. Για τη στιγμή που μιλάμε για νέες προοπτικές, διότι πέρα από το 2020 οι βιομηχανικές χώρες έχουν κάποιους στόχους σκοπεύουν να δαπανίσουν 100 δισεκατομμύρια μόνο σε αυτόν εδώ το στόχο. Θα είναι ανά, ανάλογο με την ε, βοήθεια ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να γίνει εδώ μια διάκριση. Θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση και εφιστώ την προσοχή πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή να συγκεντρωθούμε τόσο πολύ, ε, πάρα πολύ στο θέμα της μεθόδου που θα χρησιμοποιήσουμε. Επίσης να πω, υπάρχουν δύο σενάρια. Ή θα αυξήσουμε το, το πλαφόν για τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν θα το πράξουμε. Μάλλον η δεύτερη εκδοχή θα επικρατήσει, φαίνεται. Άρα να προσέξουμε να μην χάνουμε το χρόνο μας Δουλεύοντα με ένα σενάριο το οποίο δεν φαίνεται να είναι πραγματοποιήσιμο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα ήθελα να τη στιγμή που έχουμε μεικτή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των χωρών μελών θα ήταν χρήσιμο να, να κοιτάξουμε το θέμα πώς ακριβώς θα γίνει η καλύτερη χρήση ε, όσον αφορά τις συμφωνίες ανάμεσα στην Επιτροπή και τις χώρες μέλη. Είχαμε πολλές φορές είναι ευκαιρία να πούμε όταν έχουμε πόρους στις πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουμε μια φυσική καταστροφή Μπορεί, ε, δεν κάνει κανείς έλεγχο στις 27 χώρες μέλη, σίγουρα έχουν τις, πιστο, τις δυνατότητες για να αντιμετωπίσουν προβλήματα που υπάρχουν. Το ίδιο ισχύει και για την ανάπτυξη. Άρα χρειάζεται κοινό διάλογο με τι χώρε μέλη και στην, ανάμεσα στι χώρε μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλο, να πω και επιμένω σε αυτό, σήμερα το πολύ ξέρετε, έλαβα μέρο σε μια μικρή συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Θεμάτων. Αυτή η συζήτηση ήταν απογοητευτική. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Όταν μιλάμε για τον προπολογισμό εδώ πέρα υπάρχει μια συνένεση ότι πρέπει να προσέξουμε να μην ε, ξεφύγουμε φερπίνα από τα όρια. Στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων δόθηκε μια έμφαση όπου κανείς ε, έδειχνε μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο ενδεχόμενο κίνδυνο. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο όταν αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στην προσέγγιση μας. Επίσης έχουν να κάνουν με, το, ε, με την, ε, το, τον αγώνα που γίνεται κατά της, ε, της ε, ελονοσίας, της φυματίωσης. Εδώ έχει γίνει σωστή δουλειά, παραδειγματική. Αν υπήρχαν προβλήματα, εμφανίστηκαν αφότου φύγαν ήδη ή τα κονδύλια στα προγράμματα που είχαν να κάνουν με, την, ε, με αυτές τις ασθένειες. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε μια επιτροπή που δεν μπορεί να περάσει το μήνυμα. Τι μπορούμε να κάνουμε από τη δική μας πλευρά τώρα για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή ότι είναι... να συντομεύει. Ο μιλητής. Ε, εντάξει κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω εδώ πέρα. Ε, ευχαριστώ. Ο κύριος Κάσμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάντα με χαρά παρακολουθώ τον κύριο Γκέρεντ γιατί συμφωνώ συνήθως απολύτως με όσα λέει. Η η φήμη μας ολόκληρη βασίζεται στο ότι πρέπει να κάνουμε υποσχέσεις ε, που τις κάνουμε στον κατάλληλο χρόνο αλλά συνήθως αποτυχαίνουμε να τις εφαρμόσουμε ή τις εφαρμόζουμε σε λάθος χρόνο. Για μας οι αναπτυξιακοί μας στόχοι και δεσμεύσεις πρέπει να τηρηθούν γιατί έχουν υψηλή πολιτική σημασία. Γι' αυτή πιστεύουμε ότι η... το χρονοδιάγραμμα για τους στόχους της χιλιετίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρά μόνο αν βρεθούν πρόσθετα κονδύλια στο 0,7% του ΑΕΠ που έχει προβλεφθεί. Άρα το 0,7% είναι κάτι τελείως ανεπαρκές και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων των κλιματολογικών αλλαγών και της σφαιρικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε σε, που έχει πλήξει τις χώρες μας με αφάνταστο τρόπο μόνο με πρόσθετη χρηματοδότηση μπορεί να αντιμετωπιστεί. Θέλω να είμαστε οραματιστές και οραματίστριες Θέλω να εφαρμοστεί ο φόρος των συναλλαγών. Εάν ο πρόεδρος Σαρκοζή και η κυρία Μέρκελ έχουν κάτι να μας πούν σαν αυτό που είπαν στον ΟΗΕ, να το δούμε. Όταν υπάρχουν εμπορικές συναλλαγές και συναλλαγές στα χρηματιστήρια μόνο και μόνο από την εμπορία τίτλων θα έπρεπε και εκεί να υπάρξει μια φορολόγηση. Είναι και αυτός ένας πρόσθετος όρος. Δεν είμαστε βέβαια απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, ούτε είμαστε απομονωμένοι και ασύνδετοι και από τους λόγους για τους οποίους σημειώθηκε η κρίση. Το AIDS, η ελονοσία, η φυματίωση θα καταπολεμηθούν μόνο αν χορηγηθούν πρόσθετοι πόροι. Αλλά όταν μιλάμε για το 0,7% μιλάμε για το 0,7% αναπτυξιακού έτους ή κακιάς χρονιάς. Χρειάζεται λοιπόν στον τίτλο 4 μεγάλη αύξηση γιατί δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος για τη μείωση της ανέχειας στην υποσαχάρη Αφρική και την Νοτιοανατολική Ασία όταν πρέπει να αντιμετωπίσουμε απρόβλεπτες θεομηνίες όπως είδαμε τους τελευταίους μήνες. Χρειάζεται η προσθετικότητα για την αντιμετώπιση τέτοιων θεομηνιών και χρηματοπιστωτικών κρίσεων και επίσης πρέπει αν θέλουμε να έχουμε το κεφάλι ψηλά να συνδυάσουμε την αλλιευτική πολιτική και την αγροτική πολιτική γιατί φαντάζομαι ότι η παράνομη μετανάστευση και η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια θα μπορούσαν να συνδυαστούν. Άμα λυθεί το πρόβλημα της μετανάστευσης θα λυθεί κάπως και το άλλο. Με ενδιαφέρουν πολύ αυτά τα θέματα. Ξέρω ότι και εσείς έχετε το ίδιο πάθος και εσείς πρέπει να σεβαστείτε τις πραγματικότητες των προϋπολογισμών αλλά εδώ είναι η αναπτυξιακή πολιτική η επιτροπή και για μας από όλες τις ομάδες που είμαστε στην Ευρώπη οι μεγαλύτεροι δωρητές θα λέγαμε ότι αν δεν διατηρηθεί το σύστημα αυτό θα πάψουμε πια να είμαστε μια ένωση με αξίες και θα γίνουμε μια ένωση αξιών μόνο του Γκράουτσο Μάρξ. Νομίζω ότι οι αξίες μας είναι ουσιώδεις και ότι ναι, προσπαθώ να αστιευθώ αλλά δεν, δεν γελάνε από μετάφραση φαίνεται. Είναι σαν το lost in translation που λένε. Νομίζω κυρία Πρόεδρε ότι μπορώ να σταματήσω έτσι. Ευχαριστούμε κύριε Κάσμαν. Πρέπει να σας χειροκροτήσουμε για το πάθος σας για αυτά τα σημαντικά θέματα. Το λόγο έχει τώρα η Κομισιόν, η κυρία Ισαμπέλ Γκαρσόν δηλαδή. Κυρίε και κύριοι καλημέρα. Θα είμαι πολύ σύντομη. Εξετάσαμε την, το σχέδιο έκθεση ΣΥΡ με μεγάλο ενδιαφέρον θα αρκεστώ στο να αναφερθώ στην εξωτερική δράση. Σημεριζόμαστε αρκετά σχόλια από αυτά που εθίγησαν από τους μεν και τους δε. Αναμένουμε και τη θέση του Κοινοβουλίου για τα πώς θα δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος παράγων, ιδιαίτερα στα δημοσιονομικά. Αυτό σας το λέμε προς σκέψη περισσότερο ως προς τη διαφορά μεταξύ των στόχων της ανθρωπιστικής βοήθειας σε σχέση με τους στόχους και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως όλα αυτά θα μπορούσαν να εγγραφούν καλύτερα, να ενταχθούν καλύτερα σε αυτή την έκθεση. Ίσως η έκθεση ήταν ιδιαίτερα λακωνική σε ορισμένα σημεία που θίξατε ως προς τον κόσμο που ολοένα και αλλάζει. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και νομίζω ότι αυτό το σημείο που έχει ιδιάζουσα σημασία εφήγει από τον κύριο Γκέρενς αρκετά εύγλωτα έτσι ώστε να ενταχθεί στην έκθεση ΣΥΡ ακόμα καλύτερα. Και ιδιαίτερα ως προς τη συλλογική εργασία Κομισιών και Κρατών Μελών Ίσως θα μπορούσαμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι, να είσαστε πιο φιλόδοξοι από πλευράς ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό το θέμα αφορά μια γενικότερη φιλοδοξία που θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε καλύτερα σε αυτό το σχέδιο. Πρόκειται για μια εργασία σε επίπεδο 28 και όχι 27 και θα προσπαθήσουμε να το περάσουμε σε επίπεδο 27 κρατών μελών συν ενός. Μας είπατε να είμαστε πιο φιλόδοξοι, αυτό είπε η εκπρόσωπος της Επιτροπής. Να σας υποβάλω ορισμένες ερωτήσεις. Καταρχήν, η συνένεση αναπτυξιακής βοήθειας για δαπάνη 0,15% μέχρι το 2015, τότε πώς θεωρείτε θα έχει κατανομή μεταξύ των 27 κρατών μελών. Εάν αυξήσουμε το ευρωπαϊκό μέρος μέσα στα πλαίσια του 0,7%, τότε τα κράτη-μέλη θα έχουν ακόμα χαμηλότερο ποσοστό. Εάν μιλάμε όμως για αύξηση εσείς ως Κομισιόν και ως διεύθυνση υπεύθυνη για την συνεργασία και την ανάπτυξη θα έχετε την έγκριση της Επιτροπής για να κινηθούμε πέρα από την οροφή που αφορά τις δημοσιονομικές ε, προοπτικές. Γιατί αν αυξήσουμε μπορούμε να στήσουμε και το διπλασιασμό του προϋπολογισμού αν θέλουμε. Όμως μπορείτε να φανταστείτε σε τι ρήξη θα έρθετε με τους υπέρμαχους των άλλων πολιτικών. Προσπάθησα να είμαι ρεαλιστικός. Λαμβάνοντα υπόψη τις, ε, τους ε, πόρους που υπάρχουν σε επίπεδο 28 κομισιών και κρατών μελών. Και νομίζω ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε εντάχει μέσα στα πλαίσια της ε, ε, αναπτυξιακής πορείας της βοήθειας. Από τη, δύο ερωτήσεις. Από τη μια να προσπαθήσει κανείς να αναπτύξει μέσα ε, τα οποία είναι καινοτόμα για τη χρηματοδότηση εγγύηση πιστώσεων, συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και των Εθνικών Τραπεζών Ανάπτυξης και φυσικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ μπορεί κανείς να κερδίσει πολλά. Περισσότερα μπορούμε να κερδίσουμε σε μια συνεργασία ανάμεσα στις χώρες μέλη και στην Επιτροπή και μια ανακατανομή των ρόλων και των ευθυνών, εξειδίκευση και ε, που καθορίζουν ε, Επιτροπή και κράτας μέλη. Ε, η Επιτροπή, η οποία τρόπο την θα είναι το 28ο μέλο, σαν συντονιστή. Και το θέμα είναι τι θα κάνετε για να πετύχετε κάτι τέτοιο, διότι θεωρώ αν μας λέτε ότι είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι, το θέμα είναι να δούμε εσείς πώς το βλέπετε, πώς μπορούμε να πετύχουμε σε αυτήν εδώ την προσπάθεια. Ευχαριστώ, Πρόεδρος, η κυρία Κάρσον, σα ξαναδίνω το λόγο αν θέλετε να απαντήσετε στα τελευταία ερωτήματα που γίνανε. Ευχαριστώ. Σύντομα, ακριβώς υπάρχει ένα τρίγωνο ανάμεσα στο συνολικό όγκο και στον τρόπο που γίνεται η κατανομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στι χώρε μέλη, η πρόοδο που, που πρέπει να γίνει στην κοινή εργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη Χώρα μέλη. Και τρίτον, ο είπε ο κ. Μπέρμαν ότι έχουμε να κάνουμε με το, τη χρηματοδότηση και του νέου τρόπου, του καινοτόμου. Εμεί δουλεύουμε, κοιτάμε να ξαναδούμε τον κανονισμό όσον αφορά τη χρηματοδότηση, να, να δούμε σε σχέση με τα blending. Υπάρχουν κάποιε προτάσει που έχουν ήδη γίνει. Επίση, προβληματιζόμαστε να δούμε όλε τι δυνατότητε που υπάρχουν όσον αφορά το συντονισμό και τον κοινό προγραμματισμό και έχει προβλεφθεί ε, στη διάρκεια της χρονιάς κάνουν κάποιες προτάσει στην Επιτροπή και επίση στα πλαίσια του τριγώνου που σα ανέφερα υπάρχει το θέμα του υπερπολογισμού και φυσικά, φυσικά καταλαβαίνω ότι υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν Διετησίας. έχουμε τους υπεύθυνους, τους ε, πολιτικούς υπεύθυνους ε, και εδώ έχουμε να κάνουμε με το μέρος που έχει ο καθένας όσον αφορά τη βοήθεια που περνάει από, τον ευρωπαϊκό ε, προπολογισμό συγγνώμη, και εδώ έχει ε, ένα ρόλο η Επιτροπή και σύμφωνα με τους προγραμματισμούς που κάναμε εμείς έχουμε ένα 18%, 18 ε, του συνόλου της βοήθειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, 0,46 είναι η δημόσια, το ποσοστό σε, τη δημόσια συμβολή όσον αφορά την ανάπτυξη. Εμείς έχουμε στόχο να, πετύχουμε να φτάσουμε στο ύψος του 0,7% στα επόμενα πέντε χρόνια. Αν τώρα αυτή η αυξητική τάση, η απότομη, ε, μπορεί να γίνει και υπάρχει μια αύξηση του όγκου όσον αφορά τον, ε, των κονδυλίων στο ευρωπαϊκό προεκλογισμό, ε, ε, εδώ πρέπει να δούμε αν έχουμε να κάνουμε με ένα πρόβλημα ή όχι. Η θέση και η απόφαση που θα ληφθεί είναι πολιτική φύσεω. Πρόεδρο, η κυρία Χάουκ έχει το λόγο για να δευτερολογήσει. Ευχαριστώ. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στα οποία επιβάλλεται σχεδόν να απαντήσω. Αυτά που λέει η Επιτροπή Ανάπτυξη είναι ρεαλιστικά. Η Επιτροπή ΣΟΥΡ ζητάει να υπάρχουν οι απαραίτητοι πόρια. Αυτά για την πολιτική ανάπτυξη. Σε τρεις παραγράφους εμείς λάβαμε υπόψη τις ιδέες του εισηγητή. Σας το είπα, εδώ έχουμε να κάνουμε με πληρωμές που έχουν να κάνουν με τον αγώνα για τις κλιματολογικές ε, αλλαγές και εδώ είναι μια, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο, σύνοκουανών. Επίσης να πω ότι είμαστε ομόφωνοι. Πολλές φορές φυσικά κάνουμε διάλογο, συζητούμε. Ε, αλλά πολλές φορές ακούμε ότι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Ίσως, αλλά ποιος από τους συναδέλφους μου είναι πεπισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμοι να κάνουν μια επανάσταση. Όχι, όχι, επανάσταση δεν θα υπάρξει. Τουλάχιστον όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να χαιρόμαστε αν πετύχουμε σε μια αλλαγή φερπίν στη Γερμανία. Ήδη αυτό αρκεί. διότι συχνά οι επαναστάσεις οδηγούν και σε καταστροφή. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, και αυτό είναι σαφές, δεν μπορούμε να εκτεθούμε σε μια μεγάλη πίεση. Έχουμε 27 χώρες μέλη. Δεν είναι μόνο 5-6 χώρες, και ποιο πιστεύει ότι με ένα προπολογισμό ευρωπαϊκό θα μπορέσει κανεί να καταπολεμήσει, συγγνώμη, να εξαλείψει την ε, φτώχεια. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο έχει οριστεί στα πλαίσια των συνθήκων και το ανώτατο όριο 1,23% για τους ίδιους πόρους. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι με κανένα τρόπο δεν έχουμε εκ, εκμεταλλευτεί το μέγιστο κατοφλή όσον αφορεί, αφορά τους ίδιους σπόρους. Εδώ έχουμε ένα ποσοστό 1,04 και ίσως αν τα καταφέρουμε να φτάσουμε σε 1,06. Όπως είπε ο κύριος Γκέρενς, όταν συζητήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θα ενισχύσουμε τον πιλάνα για μια πολιτική ανάπτυξη, αυτό μπορεί να αποβεί σε βάρος άλλων πολιτικών. Έχουμε το θέμα το, της ανταγωνιστικότητας, ενίσχυση αυτής, ε, στην κατηγορία 3. Έχουμε τα θέματα των πληρωμών για τις εξωτερικές υποθέσεις. Και εδώ είχαμε τις πιο βασικές, τις τρεις βασικές προτεραιότητες. Τώρα αν σε αυτές τις προτεραιότητες προσθέσουμε 20% χωρίς τίποτα να αλλάξει όσον αφορά τις μεγάλες δαπάνες, κάτι που αμφισβητεί άλλος συνάδελφος, θέλω να πω ότι το 2013 βρισκόμαστε του ζώρου συνεχώ ακόμα στο θέμα του ποσοστού που είναι των ιδίων πόρων σε ένα 0,5%. Εγώ αισθάνομαι υποχρεωμένη να πω ότι η Επιτροπή, όσα, όποια και να είναι η Γενική Διεύθυνση, μας λέει καλό συνεχίστε θα μας ενισχύσει. Εδώ έχουμε να κάνουμε και τον πνευματισμό του κυρίου Μπαρόζο. Είναι αυτός ο οποίο προεδρεύει και ο οποίο θα διαμορφώσει τις μελλοντικέ κατευθυντήρες γραμμές. Τι μένει λοιπόν να κάνουμε, να ασκήσουμε πίεση στα πλαίσια της Επιτροπής. Μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. αν η Επιτροπή παρουσιάζεται μόνο όπως έχει συμβεί πολλές φορές κατά το παρελθόν σαν γραμματέα του Συμβουλίου δεν έχουμε καμιά πιθανότητα. Εμείς θέλουμε η Επιτροπή να, μας, ε, να συνεργαστεί μαζί μας, να είναι τέρος μας σε αυτή την προσπάθεια. Δεν μιλάω τώρα με την ιδιότητα του Σιωδημοκράτη εδώ για το σύνολο του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να ασκήσουμε την πίεσή μας. Θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι, τολμηροί, αλλά ε, να πω αυτό ότι δεν είναι μόνο κάτι το που αφορά τους ε, βουλευτές, αλλά έχει να κάνει με την ιδιότητα της, ε, της δυνατότητας μάλλον να κάνει κανείς νομοθετικό έργο. Έχουμε να κάνουμε μια πρωτοβουλία Αν τώρα μας λέει κάποιος ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξο, είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ θεωρώ θα πρέπει να κάνουμε ένα σοβαρό έργο και απαιτητικό. Αυτό πρέπει να γίνει από εμά. Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τις χώρες μέλη. Και όπως σας είπα πανελημένα, οι χώρες μέλη που αποτελούν το Συμβούλιο δεν είναι ένα θεσμικό όργανο της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι. Το Συμβούλιο έχει ένα άλλο ρόλο. Ενδιαφέρονται μόνο για τα δικά τους θέματα, κεφαλαιοποίηση των δικών τους θεμάτων, και τα πράγματα ήταν και παλιότερα έτσι, δεν έχουν αλλάξει. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές ε, γίνεται κανείς αυτό που λέμε μπλαζέ, αισθάνεται μια δυναμία να προχωρήσει. Θεωρώ όμως ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να απαιτήσει πόρους αρ... ικανούς για αυτή την πολιτική, να μας πούνε δηλαδή σε ένα πλάνο αυτό αυτά τα κονδύλια για, το, για την ανάπτυξη αλλά αυτό που είναι ξεκάθαρο για μας είναι ότι πρέπει να δούμε σφαιρικά το θέμα. Εμείς στη ΣΥΡ φέραμε να πετύχουμε μια συνένεση. Χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους. Νομίζω ότι έχουμε επιχειρήματα σωστά για τη βοήθεια την αναπτυξιακή. Και όλοι οι συνάδελφοι που μιλήσαν εδώ σήμερα είμαι πεπισμένη ότι θα υποστηρίξουν την Επιτροπή μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ε, παρόλο που πολλοί θα, φυσικά δεν θα θεωρήσουν ότι καλύπτονται 100% αλλά και κυρία Πρόεδρε και εγώ η ίδια δεν καλύπτομαι πλήρως από το αποτέλεσμα 100% Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ για το έργο σας. Και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο, το σημείο 6, για τον αγώνα κατά του AIDS, το... Τη φυματίωση και την ελονοσία. Το Παγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας ε, βρίσκεται εδώ για να μας μιλήσει για τα μέτρα που έλαβε σε σχέση με την κακοδιαχείριση που έχει καταγγελθεί από τέσσερις χώρες της Αφρικής ως προς τα κονδύλια του Παγκοσμίου Ταμείου και ζητήθηκε να ανασταλούν οι χρηματοδοτήσεις μέχρι το τέλος της διενέργειας της έρευνας. Επίσης, να δούμε τι θα γίνει μέσα στα πλαίσια της έκτακτης ε, Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για θέματα φυματίωσης AIDS και ελονοσίας. Δίνω το λόγο στον κύριο Εμλαντ, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα. Ο κύριος Εμπλατ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος Παγκοσμίου Ταμείου σας ευχαριστώ γιατί μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να σας δώσω ορισμένες πληροφορίες για αυτά που μάθατε από τα ΜΜΕ. Θα κάνω την παρουσίασή μου στα αγγλικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε. Ο Μπεν Ρόμπινσον, ο συνάδελφός μου, είναι υπεύθυνο για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να έχουμε αυτή την δυνατότητα, διότι θα πρέπει να έχετε πλήρη εικόνα για να γνωρίζετε πώς προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε και να ε, προλάβουμε την κακοδιαχείριση μέσα στα πλαίσια της ε, μηδενικής ανοχής. Γνωρίζετε τη δική μου θέση. Στο τέλος του Ιανουαρίου, σε ένα παραπλανητικό άρθρο του Associated Press και του επικεφαλής Ε, δημοσιεύθηκε ένα άρθρο το οποίο έπληξε ιδιαίτερα το Παγκόσμιο Ταμείο και υφιστάμεθα μεγάλες ε, πιέσεις για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το όλο θέμα ως προς τη δυσφήμισή μας. Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, οι πληροφορίες σχετίζονται με τέσσερις περιπτώσεις διαφθοράς, περιπτώσεις που το ίδιο το Παγκόσμιο Ταμείο είχε αναγνωρίσει, είχε λάβει τα σωστά ένομα μέτρα μέσα στα πλαίσια ανάκτησης των ποσών ήδη από το 2009. Άρα ε, μας καταλάβατε εξαπίνης και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από το Παγκόσμιο Ταμείο γενικότερα, διότι αυτές τις περιπτώσεις τις είχαμε ε, γνωστοποιήσει και είχαμε πει τι δράσεις θα αναλάβουμε και σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο ήδη. Μετά εκδώσαμε τις εκθέσεις μας όπου εκφράστηκε η ικανοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πλαίσια των ε, αντισταθμιστικών μέτρων και των συμπερασμάτων για το θέμα αυτό. Την έκθεση αυτή την ε, δημοσιεύσαμε στην ε, ιστοσελίδα μας και είδαμε ότι ο εν λόγω δημοσιογράφος θεώρησε ότι είχε πρόσβαση σε ένα έγγραφο εμπιστευτικού χαρακτήρα και κοινοποιούσε κάτι που δεν γνώρισαν τα εμπλεκόμενα μέρη. Όμως γνωρίζουμε ότι υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στους δωρητές μας που έχουν πολιτική μηδενικής ανοχής, κάτι στο οποίο προσβλέπουμε και εμείς και δεχόμαστε. Άρα σε μια έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο υποβλήθηκαν επιπρόσθετα μέτρα και θα πρέπει να σας μιλήσω και για το σύστημα διασφάλισης το δικό μας που ισχύει από την πρώτη μέρα της λειτουργίας μας με βάση τις δωρεές μας, όπως ισχύουν μετά το 2002. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα από αυτά τα επίπεδα διασφάλισης αφορούν την, έναν γενικό επιθεωρητή, ο οποίος μπορεί να ε, ελέγχει τα προγράμματα και οι αποκαλύψεις του ε, γίνονται, μάλλον δημοσιοποιούνται άμεσα επίσης. Έχουμε αποφασίσει να διατηρηθεί αυτή η διαφάνεια και λειτουργεί αναχαιτιστικά. Έτσι οι δωρητές μας γνωρίζουν ότι καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθούμε σε αυτό που είχαμε αρχικά ορίσει, έτσι ώστε τα χρήματα να φτάσουν στους πραγματικούς δικαιούχους. Η Γενική Επιθεώρηση και ο Γενικός Επιθεωρητής εξέφρασε την απογοήτευσή του μετά από την δημοσιοποίηση και δημοσίευση αυτή και τόνισε στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και στην Επιτροπή Ελέγχου ότι σε αντίθεση με αυτά που αναφέρονται στα άρθρα, τα προβλήματα τα οποία ήταν σοβαρά στις ε, τρεις ε, περιπτώσεις ή τέσσερις δεν αφορούν το συνολικό χαρτοφυλάκιο του Παγκοσμίου Ταμείου γιατί έγινε, μάλλον ελήφθη ένα δείγμα το οποίο δεν είναι επαρκές για να φτάσουμε σε συμπεράσματα. Ως προς τα τέσσερα επίπεδα διασφάλισης που υπάρχουν εξ αρχής. Δεν θα μπω σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά έχουμε ε, έρθει σε επαφή με διεθνείς μη κυβερνητικές φορείς των Ηνωμένων Εθνών, τοπικές μη κυβερνητικές και Υπουργεία Υγείας. Το, το πρώτο επίπεδο λοιπόν ε, αξιοπιστίας αφορά μηχανισμούς εποπτείας μέσα στα πλαίσια του βασικού δικαιούχου. Ναι. Γιατί ερχόμαστε σε επαφή αρχικά με τον βασικό δικαιούχο. Επειδή δεν έχουμε προσωπικό σε όλες τις χώρες και θα πρέπει το κόστος να παραμείνει όσο το δυνατόν χαμηλότερο, έτσι ώστε τα χρήματα αυτά να πάνε στον τελικό δικαιούχο, ερχόμαστε σε επαφή με συγκεκριμένες ε, εταιρείες ελέγχου για να πιστοποιήσουν την χορήγηση αυτών των κονδυλίων στους δικαιούχους. Πολλές φορές πρόκειται για ένα πολύ συγκεντρωτικό ε, σύστημα, δηλαδή δεν ιχνηλατούμε τη, τους δωρητές, αλλά γίνονται επιτόπιοι έλεγχοι σε τριμηνία ή εξαμηνία βάση για να δούμε τι γίνεται ε, ως προς τις ε, επιδοτήσεις αυτές. Επιπροσθέτως ζητάμε να γίνεται αιτήσιος έλεγχος του κάθε αποδόχου σε τοπικό επίπεδο και υπάρχει και το τέταρτο επίπεδο, δηλαδή μια γραμματεία η οποία ελέγχει αμφίδρομα αυτή την ε, πορεία. Και επίσης βλέπουμε τι γίνεται ως προς θέματα προμηθειών. Τέλος, και μάλλον όχι τέλος, υπάρχει το πέμπτο επίπεδο, που δεν είναι το τελικό. Και εδώ υπάρχει η βέλτιστη δυνατή πρακτική μεταξύ ε, πολυμερών, ε, μάλλον ε, φορέων πολυμερών σχέσεων όπου περίπου 30 ε, άτομα μεταφέρονται, ένα το προσωπικό αυτό μεταφέρεται σε κάθε χώρα η οποία επαληθεύει το κάθε έγγραφο. Πολλές φορές έχουμε 250.000 έγγραφα τα οποία εξετάζουμε για να είμαστε σίγουροι ως προς το που πηγαίνουν τα χρήματα. Και επίσης όλοι οι δωρητές αλλά και οι δικαιούχοι την χάνουν εποπτείας από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε, όπως σας είπα, το 2009 αρχίσαμε ε, με την ανθρωπιστική βοήθεια στη Μαυριτανία και στο τέλος του 2009 έγιναν πολλές μεταρρυθμίσεις που μετά κωδικοποιήθηκαν πέρσι τον Οκτώβριο μέσα στα πλαίσια της ατζέντα για, το για την αποδοτικότητα του Παγκοσμίου Ταμείου. Ασχολούμαστε λοιπόν με την χρηματοοικονομική εποπτεία και τους ελέγχους. Έτσι, ερχόμαστε σε επαφή με ένα ευρύτερο ε, πεδίο εντολής για επιτόπιους ελέγχους και έχουμε μία προσέγγιση αναχώρα όπου ερχόμαστε σε επαφή με τα προγράμματα προς τα πάνω. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή η συμμόρφωση, αλλά το πώς εφαρμόζονται τα προγράμματα. Επίσης υπάρχει μία ε, πολιτική διασφάλισης έτσι ώστε να γίνεται επιστροφή εξόδων και να μην προκαταβάλλονται τα έξοδα αυτά. Και ήρθαμε σε επαφή με τον Γενικό Διευθυντή για να γίνουν αγωγές εκεί που επιβάλλεται, στο Μαλί για παράδειγμα. Για το Μαλί έγινε κάτι τέτοιο. Γνωρίζουμε τις πιέσεις που αφορούν τους δωρητές μας. Υπέστην μεγάλες πιέσεις τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο έγινε μια έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου όπου ζητήθηκαν επιπρόσθετα μέτρα για τον επαναπρογραμματισμό χορηγήσεων έτσι ώστε να ενισχύσουμε τη δυνατότητα χρηματοπιστωτικού ελέγχου ως προς τον βασικό δικαιούχο να μιλήσουμε για θέματα δημοσίων προμηθειών και θα ήθελα να πω ότι έγινε ένας επαναπρογραμματισμός του 5% του προσωπικού, δηλαδή 27 προσώπων σε αυτές τις χώρες για να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος. Και προχωρήσαμε και παραπέρα έτσι ώστε να μην δούμε μόνο τους βασικούς ε, αποδέκτες, αλλά όλους τους αποδέκτες ακόμα και τους δευτερεύοντες. έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο υπάρχουν δευτερεύοντες ε, δικαιούχοι και τι χρήματα λαμβάνουν. Επίσης, γίνεται μία αναθεώρηση όλων των μηχανισμών εποπτείας και των οργανισμών εποπτείας. Θα δούνε τα δεύτερα ε, επίπεδα και θα ληφθούν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα επανόρθωσης. Ο Φέστος Μαγκάη είναι επικεφαλής που είχε συμμετάσχει στην Επιτροπή της Μποτσουάνα και στο Συμβουλευτικό ε, Συμβούλιο και ο Μάικ Λέβιτ που ε, συμμετείχε στην ε, γραμματεία από πλευράς ΗΠΑ και τουλάχιστον δύο μέλη θα προέρχονται από κράτη-μέλη για να δούμε πώς, έχουν, πώς έχει η πραγματογνωμοσύνη στον τομέα καταπολέμησης της διαφοράς. Στο μεταξύ μάθαμε ότι οι δωρητές έχουν κάπως ε, επιμεριστεί, κατακαιματιστεί. Δηλαδή έχουμε τις το τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιαπωνία, τον Καναδά, όπου ε, έχουν υπάρξει αρκετές ε, αναθεωρήσεις, δηλαδή έχουν αποχωρήσει από αυτές τις δεσμεύσεις και δεν υπάρχει καμία ανοχή για διαφθορά. Το Ηνωμένο Βασίλειο, το DFID, προέβησε μία πολυμερή έρευνα και το Παγκόσμιο Ταμείο ήταν ένα από τα εννέα, ένας από τους εννέα φορείς που είχε καλύτερα αποτελέσματα έτσι ώστε να έχουμε καινοτόμες προσεγγίσεις και διαφάνεια λειτουργίας. Και με βάση τα αποτελέσματα το Ηνωμένο Βασίλειο είπε ότι θα αυξήσει τη συνεισφορά του. Ε, κάτι το οποίο εθίγει και το οποίο χάθηκε στις ε, τελευταίες συζητήσεις είναι τα αποτελέσματα τη, του Παγκοσμίου Ταμείου. Θα μπορούσα να σας δώσω ένα διεξοδικό κατάλογο, αλλά συντηρητικά θα αναφερθώ στα προγράμματά μας 6,5 ε, εκατομμύρια ζωές έχουν ε, διασωθεί, υποστηρίξαμε 3 εκατομμύρια ε, πρόσωπα που τώρα συμμετέχουν στο πρόγραμμα καταπολέμησης HIV ενώ προηγουμένως δεν ίσχυε κάτι τέτοιο αυτό είναι πολύ σημαντικό αν δούμε πώς έχουμε δράσει τώρα τελευταία. Στην περίπτωση της ελονοσίας έχουμε μείωση της νησιμότητας άνω ε, των, ε, κάτω των 5 ετών στις χώρες που πλήττονται ενδημικά και το ίδιο αφορά και τη φυματίωση. Με βάση τα αποτελέσματά μας στο, στους στόχους της χιλιετίας μας ενδιαφέρει να δούμε ποια, ε, ποιοι πόροι είναι διαθέσιμοι και ως προς τη στοχοθέτηση του 2010 ίσως βρισκόμαστε λίγο πίσω αλλά μπορούμε να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος μέχρι το 2015. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι το 50% των πόρων μας προέρχονται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μέσα στα πλαίσια το, της ε, δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει, εάν δεν απορροφηθούν αυτά τα, αυτοί οι πόροι, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προβούμε στις ε, επιδοτήσεις, πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτές τις επιδοτήσεις. Δεν θα πρέπει να υπάρξουν καθυστερήσεις. Θα ήθελα να κάνω έκκληση έτσι ώστε να ξεπαγώσουμε όλα τα κονδύλια το συντομότερο δυνατό. Θα ήταν ε, παράλογο να γίνουν λάθη τη στιγμή που έχουν θυγεί τα κακό κείμενα και πρέπει να ενισχυθεί το σύστημά μας πριν από την ισχύ των ίδιων των άρθρων. Οι εκτελεστικοί διευθυντές θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη διαφάνεια ε, γύρω από τα εγχειρήματα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Μίτσελ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και τον κύριο Έμπλαντ για την παρουσίασή του και την παρουσία του εδώ. Είναι ένας από τους ε, δέκα καλύτερους γνώστες του θέματος και θα ήθελα να μας πει η Κομισιόν μετά από αυτά που ακούσαμε, γιατί επιμένουν στο πάγωμα των κονδυλίων. Την περασμένη εβδομάδα ακούσαμε τον Bill Gates και είπε ο, και εκείνο ότι καμιά φορά μπορεί να υπάρξει κατάχρηση κονδυλίων ή κακή χρήση. Εμείς στο Κοινοβούλιο, στην Κομισιόν, στα κράτη-μέλη Μπορεί να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει κάποια κακή χρήση κονδυλίων, αλλά στην πλειοψηφία τους τα κονδύλια χρησιμοποιούνται και στο μεγαλύτερο μέρος τους σωστά. Δεν θα ήθελα να καταδικαστούν όλοι λόγω των λαθών ορισμένων. Πάντως όσοι διαπράττουν τέτοιες απάτες βλάπτουν τους πτωχότερους κατοίκους του πλανήτη αυτό πρέπει να το ξέρουν. Οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας παραδείγματο χάρη δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς τα κατάλληλα κονδύλια. Είναι λοιπόν βασικό να ταυτιστούν και να καταπολεμηθούν και οι πιθανές ή τυχόν αυτές απάτες. Τέτοιου είδους συνοπτικές παρουσιάσεις και εκθέσεις όπως αυτή που βλέπουμε σήμερα είναι κάτι το πολύ χρήσιμο γιατί πρέπει να μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο στον δύσκολο αυτό καιρό να δεχτεί το 0,7% άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τις επιτυχίες που έχουν σημειωθεί και όχι μόνο ιστορίες για απάτες και, τε, και αποτυχίες. Λοιπόν, πρώτα το ερώτημα της Επιτροπής όταν έρθει η σειρά της γιατί παγώνουν τα κονδύλια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με όλα όσα είπε προηγουμένως ο κύριος Μίτσελ. Ευχαριστώ τον κύριο Εμπλάντ για την παρουσίασή του. Πράγματι την είχα ακούσει περίπου και σε μία από τις επιτροπές ΑΚΕ αλλά όταν διαπιστώνετε ότι μπορεί να υπάρξει λανθασμένη αναφορά, ε, έτσι είναι η πολιτική και εμείς πολλές φορές ακούμε ανακριβή πράγματα. Και όπως είπατε και εσείς, αυτά βλάπτουν, καθώς και οι απάτες, στους στοχότερους κατοίκους του πλανήτη, του πιο ευάλωτους. Ο πρόεδρος της Μποτσουάνα κάποτε είχαν ρωτήσει τον πρόεδρο της Μποζουάνα, είχαν ζητήσει από τον πρόεδρο της Μποζουάνα να κάνει μια ανεξάρτητη έρευνα για τα οικονομικά της χώρας του πράγμα το οποίο είχε θεωρηθεί τότε ως ανέκδοτο. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και σε εμά δηλαδή. Δεν είναι ίδιος ο ρυθμός απάτης, απατών που υπάρχει για όλα τα κονδύλια. Σε αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι μεγαλύτερο το ποσοστό απάτης. Πρέπει να το συγκρίνουμε με τις απάτες που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και στους δικούς τους προϋπολογισμούς για να μπορέσουμε να δούμε τη συγκριτική αξία που έχουν οι αριθμοί αυτοί. Και η παραμικρότερη δεκάρα που σπαταλιέται εδώ είναι καταστροφική. Άρα πρέπει να ξεπαγώσουν αυτά τα κονδύλια. Αν η Κομισιόν και έχω εδώ μερικές σημειώσεις για αυτά που μας είπε ο Επίτροπος Πίμπαλξ, αν η Κομισιόν θέλει να το πράξει, επειδή ανησυχεί για τις απάτες, ας κατακρατήσει ένα ποσοστό μόνο του προϋπολογισμού των προγραμμάτων αυτών, όχι το σύνολο. Ο Επίτροπος Πίμπαλξ είπε ότι θα γίνει δεύτερος δημοσιονομικός έλεγχος, ότι γίνεται αυτή τη στιγμή και ότι ως φρόνηση έχει ληφθεί αυτό το μέτρο προσωρινά του παγώματος. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται τέτοιου είδους φρόνηση. Δεν πρέπει να επηρεαστούν από τα προληπτικά αυτά μέτρα οι εφαρμογές όλων των προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί, να ξεπαγώσουν τα κοντήλια. Μέχρι το καλοκαίρι μας είπαν θα γίνει. Ναι, αλλά ίσως τότε είναι πολύ αργά. Αυτό είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε πότε ακριβώς πρόκειται να ξεπαγώσουν τα κοντήλια, για να μπορέσουμε και εμείς να δεσμευτούμε και να τιμήσουμε τις υποσχέσεις που έχουμε αναλάβει και τις δεσμεύσεις. Διότι αυτά που θα κάνουμε εμείς ως χρηματοδότηση θα τα μιμηθούν και άλλοι. Είπατε κύριε Έμπλαντ ότι ένα εκατομμύριο ειτζοπαθών έχουν στοχευθεί και ταυτιστεί. Επίσης ένα εκατομμύριο ευάλωτα παιδιά και ορφανά έχουν τύχη βοηθείας τέτοιου είδους δουλειά πρέπει να συνεχιστεί και ακόμη και για μόνο για αυτόν τον λόγο πρέπει να ξεπαγώσουν τα κονδύλια και να συνεχιστεί παράλληλα ο δημοσιονομικός έλεγχος με την πιθανότητα αργότερα μέσα στο χρόνο να ληφθούν αν χρειαστούν και πρόσθετα μέτρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρεντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε έχουμε ένα δύσκολο πρόβλημα μπροστά μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι αθώο όσον αφορά τη σοβαρότητα του προβλήματος. Μόλις παρουσιάζεται ένα πρόβλημα, πολλοί συνάδελφοι αναρωτιούνται. Η Επιτροπή δεν μπορεί να αποφύγει να ρωτήσει μια συμπληρωματική, ένα συμπληρωματικό έλεγχο. Πρέπει να το πράξει. Αυτό περιπλέκει τα πράγματα τώρα. Είναι. Ε, και εδώ ε, έχουμε μια υπερβολική απέτηση από το Κοινοβούλιο να καταλήξουμε δηλαδή στο μηδενικό ρίσκο. Όσον αφορά αυτό το θέμα, βρίσκεται σε, πρόβλημα, σε, σε, σε ένα πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με το μηδενικό ρίσκο και για τον ε, ασθενή. Εμείς δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από, το, από μικρού μας νόμους. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Να μην ε, υπερβάλλουμε, δραματοποιούμε τα πράγματα. Μου είπαν ότι το Ταμείο, το οποίο είναι αρμόδιο, ε, ε δηλαδή αυτά που είχαν προβληθεί με τον Νοέμβριο δεν θα αφορούν σε αυτό το στάδιο τους ε, ασθενείς. Έχουμε φερπίν ασθενείς από AIDS. Αν, έχουν, αν δεν έχουν πρόσβαση ε, στα κατάλληλα φάρμακα, ε, καταλήγουμε σε ένα σοβαρό πρόβλημα. Και τότε έχουμε πρόβλημα ώστε να βάλουμε τη θέση να μην μπαίνει το ρίσκο, να, μηδενικό ρίσκο εκ μέρους του ασθενούς. Η Επιτροπή μας ζητάει να προβληματιστεί μαζί μας στο να βρούμε μια λύση για αυτό το θέμα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, το Ταμείο αποκάλυψε το θέμα, διότι δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα γι' αυτό. Μέχρι την παράδοση των αντιρετροϊκών φαρμάκων. Εδώ αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση, εκτέλεση των, ε, την εκταμείευση πόρων να το δούμε με αυτούς. Διότι μόνος τρόπος είναι να αντιμετωπίσουμε το θέμα που αφορά το μηδενικό ρίσκο, κάτι το οποίο είναι υπερβολικό όπως σας είπα. Η μια άμα είναι να το σκέφτομαι έτσι, θα πρέπει να μπλοκάρουμε όλα, όλα τα κονδύλια. Δεν θα βγαίνει τίποτα. Ε, θα προσέξουμε εδώ πέρα λίγο, να μην είμαστε λαϊκιστές. Θα πρέπει να βρούμε μια λύση, να συγκεράσουμε τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε την προσοχή που απαιτεί η Επιτροπή, ε, χθε μια συνάντηση με τον Επίτροπο συζητήσαμε και είναι διατεθειμένος ο Επιτρόπος να κάνει ό,τι απαιτείται πάνω σε αυτό το θέμα. Και ευχαριστούμε την Επιτροπή αν ακορίσουμε μια μερομηνία. Διάβασα μια συνέντευξη από ένα Υπουργό για τη συνεργασία. Η διαφθορά σκοτώνει, έλεγε. να μην είμαστε υπερορθόδοξοι όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα και το ζητώ από την Επιτροπή. Να, δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία είναι κατάλληλη να βοηθήσει άμεσα και την ικανότητα να εξασφαλίσει τη χρηστή διαχείριση. Θα ήταν μια κατάλληλη θα έλεγα ε, διευθέτηση και κάτι το οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε και πολιτικά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ντέβας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα διαφθορά. Τότε γιατί η Κομισιόν πάγωσε τα κονδύλια σας. Μήπως δεν διάβασε την ίδια έκθεση με εσά. Γιατί υπάρχει αυτή η σύγχυση. Ο κύριος Έμπλαντ έχει το λόγο μετά την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ ιδιαίτερα για όσα σχόλια και ερωτήματα θέσατε πολλά από αυτά δεν αφορούσαν εμένα. Θα τα απαντήσει η Κομισιόν. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα που θα έπρεπε ίσως να τα πω καλύτερα στην παρουσίασή μου. Γίνεται αξιολόγηση επιτόπου, κάναμε ανάλυση και νομίζουμε ότι οι επιπτώσεις ε, επί των ανθρώπων που θέλουμε να ωφεληθούν και εκείνων που θα ωφεληθούν από τις δωρεές ή αντιμετωπίζουν ορισμένα τεχνικά προβλήματα για την έγκριση των χορηγήσεων. Έπειτα θα έπρεπε να είχα πει ότι κατανοούμε πλήρως την ανάγκη της Κομισιόν να συμπληρώσει, να τελειώσει τον δημοσιονομικό της έλεγχο. Εμείς συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί της με πνεύμα συνεργασίας. Οι ελεγκτές πήγαν στη Γενέβη αυτόν το μήνα, έμειναν 9 μέρες και συνεχίζουν τις έρευνές τους γιατί και εμείς έχουμε δεσμευτεί για διαφάνεια και συνεργασία με την Κομισιόν και άλλους συνεργάτες και δωρητές μας είναι δικαίωμά τους να έχουν αυτή την ασφάλεια μετά τον έλεγχο. Ωραία. Η Κομισιόν τώρα, ο κύριος Ρεγέρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία, δίνετε την ευκαιρία στην Κομισιόν να εξηγήσει τα πράγματα. Μετά τη συζήτηση που έγινε στο Κοινοβούλιο στις 16 Φεβρουαρίου, ο Επίτροπος Πίμπαλγκς είχε έρθει να σας ενημερώσει για το πώς είχαν τα πράγματα τότε. Θα ήθελα λοιπόν να εξ να πω ότι η Κομισιόν έχει συμμετάσχει πλήρως στη διαχείριση του συνολικού ταμείου με βάση την αρχή της μηδενικής ανοχής και με συνεπή τρόπο στήριξε όλες τις προσπάθειες της γραμματείας για να ενδυναμώσει, να ενισχύσει τις δυνατότητές της και πάντοτε ήταν υπέρ της επέκτασης των δικαιοδοσιών του Γενικού Επόπτη. Εμείς θεωρούμε κυρία Πρόεδρε ότι υπάρχει η εξισορρόπηση που ζήτησε ο κύριος Γκέρεντς. Έχουμε πολιτική μηδενικής ανοχής και για τις απάτες αλλά και για την στήριξη όσων τη χρειάζονται. That the, that the audit which is taking place by the Commission at this very moment. Επομένως, θα έπρεπε να πω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ο δεύτερος, το δεύτερο τμήμα του δημοσιονομικού ελέγχου που είχε αρχίσει πέρυσι όπως και άλλες διεθνείς οργανώσεις και εμείς χορηγούμε διεθνώς χρήματα και ο έλεγχος γίνεται με τρόπο πολύ ενθαρρυντικό μέχρι τώρα. Βρήκαν οι ερευνητές μερικές αδυναμίες και οι αρχές που είναι αρμόδιες για την καλή διαχείριση των δημοσιονομικών θεμάτων στο γενικότερα διαπίστωσαν και κάποια ασάφεια ως προς τις μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ χωρών. η δημοσιονομική έλεγχη και τα αποτελέσματά τους αν καταλήξουν σε κακοδιαχείριση αυτό θα σημαίνει ότι η Κομισιόν θα εφαρμόσει και επ' αυτού αυτήν την πολιτική της της μηδενικής ανοχής της κακοδιαχείρισης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι σοβαρή η κατάσταση του παγώματος των κονδυλίων και προσπαθούμε να επιταχύνουμε την ολοκλήρωση του ελέγχου. Όπως είπε και ο κύριος Εμβλάντα, είμαστε, βρισκόμαστε σε στενή συνεχή επαφή με τη γραμματεία του Global Fund και προσπαθούμε να κάνουμε τον έλεγχο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αναμένουμε τα αποτελέσματα στα τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου. Και αν είναι θετικός όπως αναμένουμε, τότε θα είμαστε σε θέση να ξεπαγώσουμε τα κανδύλια αρχές, αρχές φθινοπόρου ή τέλος καλοκαιριού. Η συνέχιση αυτή του δημοσιονομικού ελέγχου γίνεται σε απόλυτη συμφωνία με τον ανεξάρτητο δημοσιονομικό έλεγχο που αποφάσισε το Global Fund τον οποίο και, και αυτόν υποστηρίξαμε και υποβοηθήσαμε. Πάντως μπορούμε να σας δώσουμε τη διαβεβαίωση ότι αν είναι θετικός ο έλεγχος θα ξαναρχίσουν οι πληρωμές αρχές Σεπτεμβρίου και καταλήγω τονίζοντας τη δέσμευση που ανέλαβε ο Επίτροπος Πίμπαλξ εχθές στη συνεδρίαση που οργανώθηκε μαζί με τον κύριο Γκέρεντς από την οργάνωση φίλη του Global Funds Ευρώπη και όπου τονίστηκε και επενέθηκε η ταχύτητα με την οποία ανταποκρίθηκε η Κομισιόν στην κακοδιαχείριση. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι συνεχίζουμε να είμαστε δεδεσμευμένοι με το Global Fund και υπάρχει πλήρη συνεργασία και συντονισμό σε επίπεδο όλων των χωρών μελών. Ελπίζουμε έτσι να μπορέσουμε να καταλήξουμε με το πρόβλημα αυτό όσο δυνατόν γρηγορότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάτσιμαν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω ευχαριστώντας την Επιτροπή για την ειλικρινή της απάντηση και ο στόχος του, του Σεπτεμβρίου αφορά πολύ, μία περίοδο που, είναι, που αργεί πολύ. Θα πρέπει να το έχουμε λύσει μέχρι τον Ιούνιο, διότι όλοι ξέρουμε ότι αλλάζουν οι προθεσμίες. Θα πρέπει να βρείτε έναν άλλο τρόπο έτσι ώστε να, έρθουμε, να έρθετε σε επαφή και με τον Επίτροπο Πίμπαλξ για να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε εγκαίρως, διότι φοβούμε ότι ξεχνάμε τους ανθρώπους στην εμπροστοφυλακή που χρειάζονται αυτή τη βοηθεία. Γνωρίζω την ειλικρίνεια της Επιτροπής και βεβαίως ο ο, αυτός που διαβιβάζει το μήνυμα δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενό του, αλλά θα πρέπει να το θίξουμε αυτό σε επίπεδο συντονιστών. Μπορείτε να μας απαντήσετε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αν ε, δοθούν οι επιδοτήσεις μέσα στα χρονικά περιθώρια που πρέπει. Επιλύεται έτσι το πρόβλημα. Ο κύριος Ριέιρα. Θα ήθελα να τονίσω να ε, δοθεί συνέχεια στον έλεγχο αυτό και είμαι πεπισμένος Ελπίζω να μπορέσουμε να ξεπαγώσουμε τα κονδύλια. Όλα έχουν τεθεί επιτάπητος, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τη λήξη της διαδικασίας. Θα ήθελα να πω ότι η συνεισφορά της Κομισιόν στο παρελθόν δεν, έγινε, δεν ολοκληρώθηκε πριν από το τέταρτο τρίμηνο του έτους και γι' αυτό είμαστε πεπισμένοι ότι με την επιτάχυνση αυτή του ελέγχου θα ανταποκριθούμε και ο έλεγχος της Επιτροπής θα αποτελέσει παράγοντα εγγύησης για τους άλλους ε, δωρητές μέσα στα πλαίσια του ανεξαρτήτου πάνελ που θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Θα ήθελα λοιπόν εκ νέου να τονίσω και να πω ότι δεν θα πρέπει να ε, υπάρξει καμία ρήξη στο όλο εγχείρημα γιατί στο παρελθόν δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε πριν από τον Νοέμβριο. Καταβάλουμε τα κονδύλια. Ο κύριος Γκέρενς. Ε, μια ερώτηση συμπληρωματική στην Επιτροπή. Έχετε την εντύπωση μήπως ότι κάποιες χώρες μέλη που μπλοκάρανε τη συμβολή τους ε, ε αποτελούν μέρος αυτού που δημιουργείται το μπλοκάρισμα στην Επιτροπή. Μήπως έχετε μια απάντηση σε αυτό. Με συγχωρείτε που παρεμβαίνω, αλλά πολύ πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε μία συνάντηση με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκοσμίου Ταμείου σε, στην περίπτωση ορισμένων χωρών θεωρήθηκε ότι δεν ήταν σε θέση ήδη να δεσμευτούν στην σύσκεψη της Νέας Υόρκης. Άρα αυτές οι χώρες, οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα περιμένουν τα αποτελέσματα του ανεξάρτητου πάνελ που θα φτάσουν αργότερα. Το ζήτημα είναι ότι εάν επέμβουμε τον Ιούνιο, Ιούλιο και αν έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σε σχέση με το ανεξάρτητο πάνελ, τότε θα αλλάξουν τα δεδομένα και όταν έχουμε τα τελικά αποτελέσματα του πάνελ θα μπορέσουμε έγκαιρα να παρέμβουμε και με βάση τα νέα δεδομένα. Ο κύριος Εμπλάντ. Προσπαθώ να δω από τις ε, σημειώσεις μου που πρέπει να απαντήσω. Ο κύριος Μίτσελ αναφέρθηκε σε ορισμένα θέματα, αλλά εσείς αναφερθήκατε σε θέματα που αφορούν αμεσότερα την ε, Κομισιόν. Είπατε ότι δεν θέλετε πια να ακούσετε για ε, διαφθορά. μπορείτε να δεχτείτε αυτά που είπε η Κομισιόν και οι περιπτώσεις διαφθοράς ήταν γύρω στις 8-9. Το Ηνωμένο Βασίλειο ασχολήθηκε, σε, ασχολήθηκε με 30 υποθέσεις και είμαστε ή σε, περίοδο, σε δοκιμαστική περίοδο ή μειώνονται τα κονδύλια. Αυτά αναφέρονται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχαμε να κάνουμε με 10 ε, πολυμερείς και οι 8 έχουν μπει στην υψηλότερη κατηγορία. Τα καταφέραμε πολύ καλά ως προς τη σχέση κόστους-οφέλους με βάση και την κατάσταση των δωρητών και ως προς το δεύτερο ερώτημά σας, εάν μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με αυτό το χρονοδιάγραμμα, θα είμαστε πολύ καλά αν και οι άλλοι δωρητές μπορέσουν να ακολουθήσουν αυτό το χρονοδιάγραμμα. Δεν λέω ότι οι δωρητές, υπάρχουν δωρητές που κρύβονται πριν πίσω από την Επιτροπή, αλλά ένας μεγάλος δωρητής όπως η Κομισιόν που έχει το, την επαγγελματική πείρα και το προσωπικό σε σχέση με μικρότερους δωρητές, οπωσδήποτε θα αποτελέσει σηματοδότη για τη μελλοντική κατάσταση. Τώρα, επειδή έχω ασχοληθεί με πολυμερή στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, θεωρώ ότι οι εσωτερικοί μηχανισμοί έχουν βελτιωθεί έτσι ώστε να μην χρειάζεται οι υπογράφοντες να περιφέρονται σε γραφεία της Κομισιόν από τη μια άκρη στην άλλη. Και ο κύριος ε, Κάσμαν, ίσως υπάρχουν ολιστήσεις και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει διαρκής έλεγχος. Ως προς τα σχόλια άλλων μελών, συμφωνώ με άλλα αποτελέσματα και συμπεράσματα τον κύριο Κάσμαν έτσι ώστε να μην υπάρχει μεταβίβαση του ιού από τη μητέρα στο παιδί. Μιλήσαμε για ε, παρακράτηση μιας ποσοστίας αναλογίας. Δεν αυτός δικός μου ρόλος, αλλά είδαμε μία ανταπόκριση η οποία δεν ισχύει και για τους δικούς μας ε, αποδέκτες. Δηλαδή προσπαθούμε να προστατεύσουμε το σε μέρος του προγραμματός μας μέσα στα πλαίσια της ε, μηδενικής ανοχής για, την, ε, για το σφετερισμό ή κακοδιαχείριση. Ως προς την έκθεση DFID, ήταν ένα εγχείρημα όταν ε, ανήλθε στην κυβέρνηση παρούσα, ε, ανέλαβε μάλλον η παρούσα κυβέρνηση. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτούς τους δωρητές. Το 2009 άρχισε η διαδικασία ελέγχου. Λάβαμε αυτή την ε, έκθεση αρκετά αργά το 2010 και χαιρόμαστε για το follow-up γιατί προχωρήσαμε αρκετά. Σας ευχαριστώ και πάλι, Πρόεδρε, και την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Σας ευχαριστώ που παρευρεθήκατε εδώ και μας δώσατε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε. Το επόμενο θέμα, θέμα στην ημερήσια διάταξη, καταπολέμηση της παράνομης ηλίας σε παγκόσμιο επίπεδο, Έχουμε τον συνάδελφο που έκανε μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή Αλίας, ο κ. Ποντός λοιπόν ο οποίο έκανε αυτή τη γνωμοδότηση, θα πάρει και το λόγο στην αρχή. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, με λίγες λέξεις θα παρουσιάσω τη γνωμοδότηση που συνέταξα για την Επιτροπή Αλίας για τον αγώνα της καταπολώνησης τη παράνομης Αλίας σε παγκόσμιο επίπεδο και το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Έδωσα έμφαση στο θέμα της ανάπτυξη. Τέσσερα σημεία θα πρέπει να, να τα υπογραμμίσουμε, έτσι μου φαίνεται. Είναι σημαντικό να δούμε τη σχέση ανάμεσα σε μια νόμιμη προγραμματισμένη αλία για την οικονομική ανάπτυξη, πράσινη, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στι αναπτυσσόμενες χώρες οι συνέπειες τη παράνομη αλληλεία είναι μεγάλες για το περιβάλλον αλλά και για την οικονομία. Ακόμα περισσότερο στις χώρες τι αναπτυσσόμενε. Η παράνομη αλληλεία πλήττει την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, γίνεται κατάχρηση των πόρων και θέτει σε κίνδυνα τα αποθέματα ηχθείων. Επίσης να επενθυμίσω ότι ο αγώνας αυτός είναι κάτι που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Απαιτεί συμφορι... σφαιρικές λύσεις και από όλες τις χώρες μέλη. Μου φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια ανικανότητα τεχνική όσον αφορά τις χώρες μέλη και στις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε να επιβάλλουμε τις ίδιες περιορισμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις ανεπτυγμένες. Όπως υπογραμμίσει επανειλημμένα στην Επιτροπή μας, Ορισμένες νησιωτικές χώρες, το τομέα Φερρυπίν, έχουν περιορισμένες ικανότητες. Θα πρέπει λοιπόν να τις ε, βοηθήσουμε σε αυτόν τον αγώνα κατά της παράνομης αλίας. Γι' αυτό έδωσα έμφαση όσον αφορά την ενήγηση την χρηματική σε αυτόν τον τομέα όταν κάνει συμφωνίες η Ευρωπαϊκή Ένωση με χώρες αναπτυσσόμενες. Επίσης υπάρχει αναγκαιότητα για μια πολιτική συνεκτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνέπεια με όλε τι πολιτικέ και το επιθυμεί συνεχώ η Επιτροπή μα. Αυτό πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Και τέταρτον, στην εφαρμογή ε, τη κοινωνία των πολιτών και να γίνει εδώ να συμβάλλουμε στον αγώνα κατά της παράνομης αλίας. Μια σφαιρική λοιπόν προσέγγιση όσον αφορά αυτό το θέμα. Κατάσταση των πρωτοπολιών στις 19 Απριλίου στις 12 η ώρα. Είμαι στη διάθεσή σας και ευχαρίστω να ακούσω τα οποιαδήποτε σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και Λοιπόν, το λόγο θα πάρει η Επιτροπή για κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τις παρατηρήσεις την εισαγωγή που έκανε ο κ. Πόγκα έχω εδώ πέρα εκ μέρους της Επιτροπής. Η Επιτροπή επιθυμεί να πάρει το λόγο ή όχι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να σχολιάσουμε επί του παρόντος. Θα θέλαμε όμως να τονίσουμε ότι αυτό το έγγραφο εργασίας την χάνη της υποστήριξης της Επιτροπής θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την παράνομη αλίευση, θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους πάντες Νομίζω ότι μιλάμε και για οργανωμένο έγκλημα. Και πολλές φορές έχουμε να κάνουμε με υπηκόους τρίτων χωρών που ε, ζουν σε μια τέταρτη χώρα. Θα επανέλθουμε για σχόλια αργότερα. Euh, Ευχαριστώ. Είναι ενδιαφέρον αυτό που μας είπατε. Είναι και τα θέματα που αφορούν την Επιτροπή μας, δηλαδή την, ε, το ξέφλυμα χρήματος σε φορολογικούς παράδεισους. Είναι ένας συνεχόμενος αγώνας και αφορά και αυτός αγώνας στην Αλία. Τώρα, στο 8 περνάμε τις για τον κανονισμό 1905 του 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης αναπτυξίας αναπτυξιακής συνεργασίας, ποια είναι τα διδάγματα και οι προπτικές για το μέλλον. Η Επιτροπή μας αποφάσισε να είναι δραστήρια όσον αφορά αυτό το μηχανισμό. Έχουμε τον συνάδελφό μας κύριο Μίτσελ και είναι σημαντικό να συζητήσουμε σε αυτό το στάδιο τις θέσεις μας όσον αφορά το μηχανισμό ούτω ώστε το που θα διαδεχθεί το DCI. Οι επιπτώσεις θα υπάρχουν ε, και στο χρηματοδότηση για την πολιτική ανάπτυξη για το μετά το 2013. Η, η έκθεση του κυρίου Μίτσελ λοιπόν είναι πολύ σημαντική για ένα πιο ευρύ διάλογο για τα, στα πλαίσια ενός ε, προγράμματος ε, πολιετούς για τη χρηματοδότηση και έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να τροφοδοτήσει αυτό το διάλογο. Κύριε Μίτσελ, έχετε το λόγο. Um, <clears throat> uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η προηγούμενη συζήτηση για τη μελλοντική χρηματοδότηση της Ένωσης και τη δουλειά της Επιτροπής ΣΟΥΡ αποσαφήνισε ότι χρειάζεται επαρκή επαρκής χρηματοδότηση στο πολιετές καινούριο πλαίσιο. Γιατί οι πόροι για τις εξωτερικές δράσεις θα παραμείνουν χαμηλοί, ενώ τα προγράμματα παράλληλα είναι πολλά. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποια διασφάλιση ότι τα χρήματα που θεατεθούν θα δαπανηθούν με τρόπο αποτελεσματικό και συνοπτικό ώστε να εξυπηρετεί πράγματι εκείνους που θέλουμε να ωφεληθούν. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε την αρχιτεκτονική και την ομοθεσία που διέπουν ε, τα αναπτυξιακά προγράμματα. Στο σχέδιο έκθεσής μου προσπαθώ να ορίσω ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι μας με βάση τα μαθήματα που πήραμε από το παρελθόν. Ελπίζω να συμφωνήσουμε για τις βασικότερες αρχές που θα αποτελέσουν τις βάσεις για τις διαπραγματεύσεις που θα, γίνουν, θα αρχίσουν φέτος. Θα σας πω λοιπόν τις βασικές αρχές για την επόμενη αναπτυξιακή πολιτική. Βασικά χρειάζεται ένας μηχανισμός της συνεργασίας που να στοχεύει ειδικά τις αναπτυσσόμενες χώρες για, με στόχο τη μείωση και κατάργηση της ανέχειας. Το νέο αυτό εργαλείο ημέσων πρέπει να βασίζεται, να στοχεύει ιδιαίτερε φτωχότερε χάρη και φτωχότερε περιφέρειε των χωρών για να χρηματοδοτηθούν μέτρα που θα πληρούν τα κριτήρια για βιώσιμη ανάπτυξη όπως την ορίζει ο ΣΑΧ. πρέπει η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια να είναι τουλάχιστον όσο αποτελεσματική ήταν και στο προηγούμενο πρόγραμμα, στο μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας. Τέτοιου είδους συνεργασία πρέπει να χορηγείται από χωριστά εργαλεία για να προστατευθούν οι ιδιαιτερότητες της αναπτυξιακής συνεργασίας η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και η μη επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια είχαν συνδυαστεί με τρόπο που δεν μπορούσαμε να ταυτίσουμε ακριβώς. Αυτό θα αλλάξει στο μέλλον. Το νέο εργαλείο επίσης θα εφαρμόζεται και στις χώρες μας και στις χώρες που όρισε ο ΣΑ. Δηλαδή πρώτα πρέπει να δούμε τι είναι αναπτυσσόμενη χώρα Υπάρχουν σοβαροί λόγοι να συνεχιστεί επίσης η χορήγηση βοήθειας και σε χώρες μέσου εισοδήματος. Βασικές δραστηριότητες όπως οι υγειονομικές ας πούμε θα βασίζονται στις διεθνείς αρχές, δηλαδή τουλάχιστον 20% της χρηματοδότησης για τα γεωγραφικά προγράμματα θα αφιερωθεί σε αυτά. Τέλος, το νέο εργαλείο πρέπει να έχει αρκετή χρηματοδότηση και να μην μειωθεί σε σύγκριση με το τωρινό, αλλά να αυξηθεί μάλιστα. Γιατί η βοήθεια της Ένωσης είναι ιδιαίτερη. Συντονίζει αυτά που λέει το άρθρο 210 της Συνθήκης Λισαβόνας και ο προϋπολογισμός της Ένωσης συμμετέχει στην επίτευξη του στόχου του 0,9%. Τα οι τελευταίοι αριθμοί λένε ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ανέρχεται αυτή τη... θα χρειαστεί 10 δισεκατομμύρια για να επιτύχει ο στόχος που έχουμε θέσει λόγω του περιορισμού που πρέπει να σεβαστώ στο μήκος της εκθεσής μου Χρειάστηκε να περιορίσω και αυτά που ήθελα να συμπεριλάβω στους στόχους με θέματα όπως τη συνεργασία με περιφερειακές και τοπικές αρχές και θα ήθελα να καλέσω την Κομισιόν για μακροοικονομικά θέματα όπως την ανάπτυξη επιχειρησιακού πνεύματος να προβλέψει κάτι για την επιμόρφωση στους τομείς αυτούς στις αναπτυσσόμενες χώρες με βάση την εμπειρία της Επιτροπής μας και των ομάδων εργασίας για τον δημοκρατικό έλεγχο του μηχανισμού χρηματοδότησης της έχουμε δει ότι και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν έχουν ωφεληθεί και μας έδειξαν οι μελέτες μας αυτές ότι μπορεί να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα τα οποία στο μέλλον μπορούν να αποφευχθούν. Ιδιαίτερα είδαμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος, ο στόχος της εξάλληψης της ανέχειας να επισκιαστεί από άλλα συμφέροντα και θέματα. Κυρία Πρόεδρε, μετά τη θέση της συνθήκης της Λισαβόνας δεν αρκεί πια ο ισχύων μηχανισμός χρηματοδότησης. Πρέπει το Κοινοβούλιο ε, σε ισοδύ... με ισοδύναμο τρόπο με το Συμβούλιο να συμμετέχει στη λήψη των βασικών αποφάσεων για αυτά τα θέματα. Όπως ξέρετε, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας για το μέλλον και αναμένω τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστούμε πολύ. Η Κομισιόν, η κυρία Γκαρσόν. Σας ευχαριστώ και πάλι. Θα πρέπει να πω ότι καλωσορίζουμε και χαιρόμαστε για τα νέα δεδομένα της έκθεσης Μίτσελ. Πολλά ουσιώδη σχόλια αναφέρθηκαν θα ήθελα να αναφερθώ στο 0,7% τον απότερο στόχο για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και εμείς αυτό έχουμε θέσει ως όριο σε επίπεδο προϋπολογισμού και για να καλύψουμε μεταξύ άλλων το μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας. Είμαστε της άποψης ότι το μέσο αυτό αναπτυξιακής συνεργασίας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τα νέα αυτά δεδομένα ως προς μια ενδεχόμενη διαφοροποίηση δράσης σύμφωνα με διαφορετικούς στόχους όπως αμοιβαίο συμφέρον και ούτω καθεξής. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες εναλλακτικές και λαμβάνουμε υπόψη τα δεδομένα του εισηγητή. Επίσης, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο, στους στόχους εκπλήρωση των αναπτυξιακών, στό, αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Ίσως χρειάζεται κάποια διαφοροποίηση πίση μεταξύ δικαιούχων χωρών και διαμόρφωση της ενίσχυσης για στοχοθέτηση στις ε, φτωχότερες χώρες, ενώ να προωθήσουμε διαφορετική συνεργασία με αναδυόμενες χώρες. Επίσης λαμβάνουμε υπόψη τα σχόλια ως προς τα θεματικά προγράμματα και θα θέλαμε να πούμε ότι σε αυτό το στάδιο προσπαθούμε να δούμε πώς θα θέσουμε στόχους με βάση τις νέες παγκόσμιες προκλήσεις και ποιος είναι ο καλύτερος θεματικός στόχος μέσα στα πλαίσια της αλληλεγγύης και συμπληρωματικότητας της περιφερειακής συνεργασίας. Επίσης, συμφωνώ με την έκκληση για καλύτερο συντονισμό μεταξύ Κομισιών και κρατών μελών και να επιβεβαιώσω και τη θέλησή μας να βελτιώσουμε το διάλογο μεταξύ Κομισιών και Κοινωνίας των Πολιτών συμπεριλαμβάνοντας και τον ε, διαρθρωμένο διάλογο ο οποίος έχει προωθηθεί και προωθείται εδώ και ένα χρόνο με την κοινωνία των πολιτών. Uh, Έτσι ώστε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε αυτά τα δεδομένα κατά το καλύτερο δυνατόν στα, στα, στις μελλοντικές μας επιδόσεις και προγράμματα. Θα ήθελα επίσης να πω ότι, καλ, ότι καλωσορίζουμε την ιδέα ευφυούς ευελιξίας στον τρόπο προγραμματισμού της βοήθειας και να πω ότι θα πρέπει να εισαγάγουμε μερικές από τις καλύτερες πρακτικές του Ταμείου Αναπτυξιακής Βοήθειας για να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε το μηχανισμό αναπτυξιακής βοήθειας. Mm. Τέλος, στην έκθεση μιλάμε για θεματικά προγράμματα για τη μετανάστευση και τη χορήγηση ασύλου. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι μέχρι τούτε το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης έχει τύχει ελέγχου. Uh, a, point on that. Um, as regards the, recommendation made for the... Αφορούσε την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Άρα, τα θεματικά προγράμματα θα πρέπει να συμπληρώνουν της δράσεις σε επίπεδο χώρας, που είναι και το βασικό επίπεδο συνεργασίας. Άρα δεν συμφωνούμε απόλυτα με αυτά που προβλέπονται ως προς επενδύσεις. Εάν σημαίνει ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας αφορούν μόνο το κρατικό επίπεδο. Ίσως εμείς δεν κατανοούμε καλά το κείμενο, αλλά θεωρούμε ότι η δράση ως προς αναπτυξιακούς στόχους εμπίπτει σε κρατικά προγράμματα. Εκεί υπάρχει καλύτερη διάδραση με τις χώρες και ε, είναι και η καλύτερη επένδυση, ο καλύτερος τρόπος επένδυσης, αλλά ίσως αυτό αποτελεί μία παρανόηση από δικής μας πλευράς. Ας σταματήσω εδώ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έκθεση. Εντάχει, λέει ο κύριος ε, Μίτσελ, υπάρχει γενικά συμφωνία σε μερικούς τομείς ε, θα πρέπει να ε, καταπραίνουμε ορισμένα, ορισμένες διαφορές ή διαφωνίες ως προς το ιδιοκτησιακό και το ε, επιχειρηματικό πνεύμα που μας ε, ε, διέπει ως προς τη βασική εκπαίδευση ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μία άλλη προσέγγιση. Δηλαδή, εάν ο καθένας έχει τα μέσα, τότε μπορεί να αντεπεξέλθει. Όταν μεταβαίνουμε στην Αφρική, Υπάρχουν ε, μεγάλοι και μακρύ, μακρύς κατάλογοι και πολλές φορές όταν μεταβεί κανείς στην ε, Αφρική βλέπει ότι υπάρχουν ε, κινητά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ καλύτερα από το δικό μου κινητό. Ο συνάδελφος Ντέβα μίλησε για υπολογιστές που μπορούν να κινηθούν με την ηλιακή ενέργεια αποκλειστικά. Άρα δεν θα πρέπει να δούμε την εκπαίδευση στρίκτο σένσου, αλλά να δούμε την εκπαίδευση ως μέσον πλούτου. Και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη από την ομάδα. Δηλαδή, εάν μπορέσουμε να λύσουμε κάπως το ιδιοκτησιακό καθεστώς θα μπορέσουμε να δούμε και θέματα νέων ευκαιριών. Στον τομέα της επιστήμης των επιστημών υπάρχουν νέες δυνατότητες. Στη Νότια Αφρική και στην Αυστραλία υπάρχουν νέα σχέδια και για την Αφρική θα ήταν πολύ, ιδιαίτερα για την Αφρική θα ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί όταν κάποιος ε, καίγεται δεν μπορούμε να πούμε ότι χτίζουμε μία πυροσβεστική και να δώσουμε αυτή την απάντηση. Αλλά μπορούμε, μπορούμε να έχουμε μία μονάδα πρώτων βοηθειών. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Έτσι θα πρέπει να διαχειριστούμε και κατά τον καλύτερο τρόπο τα χρήματα που έχουμε. Στις 13 Απριλίου στις 4 το απόγευμα είναι η προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών. Σημείο 9 της σημερινής διάταξης. Κύριος Σφένσον, γνωμοδότηση για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα εκδημοκρατισμού. Ε, Ορίστε κύριε Σφένσον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από έξι χρόνια η Κοντολέζα Ράις έκανε μια ομιλία στο Κάιρο, πολύ χαρακτηριστική. Έχουμε εξασφαλίσει σταθερότητα εις βάρος της δημοκρατίας στην Μέση Ανατολή. Είναι σαφές ότι η Δύση ήταν πολύ ικανοποιημένη με τη σταθερότητα. Είχαμε αυθαίρετες ηγεσίες οι οποίες δεν δέχτηκαν πιέσεις για να βοηθήσουν την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή την δημοκρατία. Πριν από δύο χρόνια, στην συνάντηση τη, στην Ιταλία της ομάδας των Οκτώ, ακούσανε ε, τον Καντάφη και τώρα διαπιστώνουμε ότι στη Λιβύη οι νέοι είναι διατεθειμένοι να χάσουν τη ζωή τους για να καταπολεμήσουν τη δικτατορία. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι στο μέλλον η δημοκρατία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Αυτός ο οποίος περιμένει να υπάρχει διαρκής ε, σταθερότητα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στη δημοκρατία. Ε, το θέμα της δημοκρατίας είναι επίκαιρο μεγάλο μέρη, μεγάλα μέρη στον κόσμο ε, ε αναπνέουν, προσδοκούν να δουν μια δημοκρατική εξέλιξη. Και εδώ υπάρχει θέμα ευθύνη. Το θέμα της δημοκρατίας δεν είχε να κάνει μόνο με ελεύθερες εκλογές. Ξέρουμε ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω για να έχουμε μια, ένα πολιτισμό δημοκρατίας, ένα πλαίσιο δημοκρατίας. Χρειάζεται κάτι παραπάνω από τις ελεύθερες εκλογές. Η ελευθερία έκφρασης ε, και θα πρέπει να μπορούν να αναπτυχθούν οι ιδέες και να εκφράζεται κανείς χωρίς να ελέγχεται από το κράτος. Το θέμα όμως της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα δημοκρατισμού μας ανισχύει διότι υπάρχει μια πολιτικοποίηση αυτού του θέματος. Υπάρχει το θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ε, κυριαρχία των ε, κρατών, λένε μερικοί. Εγώ δεν συμφωνώ απολύτω με αυτού. Βρισκόμαστε σε ένα αποφασιστικό σημείο για την εξέλιξη στον κόσμο. Και είναι σαφέστερα, σαφέστατα ότι σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβάλλει, να βοηθήσει τα δημοκρατικά κινήματα και τα νέα και τα πολιτικά κόμματα στι νέε δημοκρατίε. Το θέμα του εκδημοκρατισμού δεν έχει να κάνει μόνο με την ομανιστική πτυχή, αλλά είναι και καθήκον μας σε σχέση με τη συνθήκη. Ε, δεν έχει να κάνει εδώ πέρα το θέμα αυτό που λένε πολύ πολιτιστικό υπεριαλισμό. Έχουμε Αυγανές οι οποίες μισούνε, συχαίνονται τους Ταλιμπάν. Έχουμε στην Κίνα περιπτώσεις, έχουμε διάφορα μέρη του κόσμου. ο Σαντάμ Χουσέιν ε, τρομοκρατούσε το κόσμο του, το λαού του. Το θέμα της δημοκρατίας δηλαδή δεν είναι κάτι που το έχουμε ε, εμπνευσεί, δημιουργήσει εδώ στην Δύση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με αξίες οι οποίες είναι οικουμενικές θα λέγαμε και ισχύουν για τον κάθε άνθρωπο. Και αυτό ισχύει σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλες τις υπήρους. Κύριε Πρόεδρε, όταν μιλάμε για δημοκρατία, αυτό είναι η ψυχή του προβλήματος. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με κάθε άτομο, την αξιοπρέπεια αυτού. Η δημοκρατία χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται υπομονή. Αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι η διαδικασία αυτή σταματάει, φρενάρεται. Η δημοκρατία και οι ανθρώπινες αξίες θα πρέπει να μην διαχωρίζονται. Δεν μπορούν κατ' εμέ. Σίγουρα υπάρχουν πολλές πτυχές όσον αφορά την ανάπτυξη, τον εκδημοκρατισμό και τη βοήθεια που μπορεί κανεί να δώσει. Εγώ έχω μια, μια μικρή γνωμοδότηση, είναι μικρή ίσω, αλλά είμαι ανοιχτό, δέχομαι τη, δική σας, ε, ε, τη δική σα συμβολή και είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Θέλει κανείς το λόγο. Μάλιστα. Ο κύριος Βίσας. Φίσας. Ναι, ορίστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ενημερώσω την Επιτροπή για τις τελευταίες εκλογές. Α, συγγνώμη. Ε, δεν κατάλαβα καλά. Συγγνώμη, συγγνώμη. Μιλάμε για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εκδημοκρατισμό. Η κυρία Σαμπόρσκα, μήπως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφό μας Σβένσον για τη γνωμοδότησή του. Νομίζω ότι πέφτει σε πολύ κατάλληλη χρονική στιγμή. Εδώ και πέντε μήνες είχαμε πρώτο σκεφτεί να γίνει αυτή η γνωμοδότηση και τελικά είμαστε ικανοποιημένοι στα πλαίσια της τωρινής συγκυρίας. Ο κ. Σβένσον μίλησε για κοινωνικά κινήματα, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, πολιτικά κόμματα. Πιστεύω ότι πρέπει να αναφέρουμε και τις γυναίκες να δώσουμε δηλαδή ειδική έμφαση στις γυναίκες ως τους ανθρώπους που φροντίζουν άλλους και πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να αρχίσει διάλογο με δημοκρατικά όργανα όπου επικεφαλής υπάρχουν γυναίκες και να ζητήσουμε να τις καλέσουμε να μας βοηθήσουν γιατί πολύ λίγοι γνωρίζουν καλύτερα από αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε μη δημοκρατικές χώρες όπως η κυρία Ντεκάιζερ που έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα εδώ και πολύ καιρό. Έχω πάει και εγώ σε διασκέψεις για το θέμα αυτό όπου είχε συζητηθεί γιατί οι γυναίκες είναι πάντα στην πρώτη γραμμή του εκδημοκρατισμού η απάντηση που δίναν οι γυναίκες επιτόπου ήταν ότι εκείνες βλέπουν το πρόβλημα και μέσα από τα μάτια της οικογένειάς τους, των παιδιών τους, των αντρών τους που βρίσκονται ίσως εκείνοι στην πρώτη γραμμή των μαχών. Άρα οι γυναίκες είναι σίγουρο ότι βρίσκονται, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες εκδημοκρατισμού και γι' αυτό θα ήθελα να υποβάλω μία τροπολογία μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει προβλεφθεί όπου να μιλήσω και για τις γυναίκες. Η κυρία Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ δεν είμαι η σοσιαλιστή Σκιώδης αλλά η Σκιώδης επί της ουσίας στην ΕΠΕΞ και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω την απόψή μου. Ξημερίζομαι σχεδόν απόλυτα όλα όσα είπε ο κύριος Σφέντσον. Εξάλλου και η έκθεσή μου κατά πρώτο λόγο για τέτοιου είδους αλλαγές μιλάει. Σίγουρα κάναμε λάθος όταν βάζαμε σαν πρώτη στο στόχο τη σταθερότητα ενώ έπρεπε να είναι η δημοκρατία. Συμμερίζομαι επίσης την άποψη που εκφράσατε ότι δηλαδή σε αυτές τις δικασίες εκδημοκρατισμού έχουν μια πολιτική διάσταση την οποία δεν βλέπουν στο σύνολό τους οι διάφορες αποστολές παρατήρησης κτλ. Όλα αυτά τα είχα πει και εγώ, θα δω αν υπάρχουν επικαλύψεις ή όχι, αλλά πάντως είμαι υπέρ αυτών που είπατε. Το ίδιο ισχύει για την ελευθεροτυπία, τα νέα μέσα ενημέρωση κτλ. καθώς και Συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Ζαμπόσκα για το ρόλο των γυναικών στον εκδημοκρατισμό. Εκεί όπου δεν μίλησα πολύ στην έκθεσή μου, το θέμα για το οποίο δεν μίλησα πολύ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ καιρό θεωρούσε ότι η δημοκρατία ή μη στις χώρες με τις οποίες συνάπτε συμφωνίες ήταν δευτερεύον θέμα σε σύγκριση με τη σταθερότητα, αλλά δεν αρκεί. Αυτό πρέπει τώρα να δώσουμε πολύ πιο πολιτική διάσταση σε όλα αυτά. Αυτό δεν το επανέλαβα ίσως επαρκώς ε, και στα πλαίσια της ανάπτυξης γιατί δεν θα ήθελα ο εκδημοκρατισμός να είναι και αυτός μόνο πολιτικός. Οι αραβικές εξεγέρσεις σήμερα το δείχνουν Υπάρχει μία πολιτικο-οικονομική αλληλεξάρτηση. Θέλουμε να είναι τα πράγματα να τα δούμε πολύ πιο πολιτικά, να μιλάμε πολύ περισσότερο για τη δημοκρατία, αλλά και για σημαντική στήριξη των κοινωνικο-οικονομικών πτυχών. Αν λοιπόν στην έκθεσή σας κύριε Σβένσον, στην ομοδότησή σας, αλλάξετε τι τίποτα, θα ήθελα να μην ξεχάσετε αυτά που ανέφερα. Αύριο το μεσημέρι λίγη η διορία κατάθεση τροπολογιών και θα ήθελα γενικά να πω ότι βρισκόμαστε στην ίδια γραμμή. Ο κύριος Μίτσελ. Ναι, και εγώ δέχομαι την έκθεση αυτή. Είναι πολύ επίκαιρη, το είπε και η κυρία Ζαμπόρσκα. Ιδιαίτερα θα ήθελα να τονίσω το σημείο τα και να πω ότι καιρό είναι πια να ξαναδούμε τις σχέσεις μας με ορισμένες χώρες. Στη Βόρεια Αφρική ας πούμε δεν δέσποζε δεν ε, κυριάρχησε η δράση των πολιτικών, δεν έσπρωξε αυτή τον κόσμο αλλά η πρόσβαση στο διαδίκτυο και τέτοια πράγματα. Όταν δοθεί η ευκαιρία δηλαδή ο κόσμος εξηγίζεται. Οι δικτάτορες που ανατράπηκαν εκεί δεν είναι οι μόνοι και Ε, στη Βόρεια Αφρική είδαμε μεγάλη αλληλεγγύη και μεταξύ των ανθρώπων εκεί, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τις σχέσεις μας με άλλους δικτάτορες. Πολύ επίκαιρη πάντως η έκθεση και συγχαίρω τον κύριο Σιβένσον. Ο κύριος Γκερέρος Αλάμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βρισκόμαστε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Υπάρχει, υπάρχει ένας εισηγητής επί και ένας ε, ε Θα πρέπει να πάρουμε θέση και στις δύο περιπτώσεις. Θα ήθελα να πω εγώ το εξής, ότι όσον αφορά τον εκδημοκρατισμό θεωρώ είναι μια μοναδική εποχή την οποία ζούμε Είδαμε ένα τρίτο κύμα εκδημοκρατισμού Φερρυπίν μετά. Είχαμε δει ε, τις φάσεις της ευρωπαϊκές, τώρα βλέπουμε ε, μια νέα περίπτωση με ένα νέο κύμα, μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση όπου βλέπουμε ότι μετά από τις φάσεις του που είδαμε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο είναι σε μια Ήπειρο όπου δεν υπήρχε παράδοση δημοκρατική. Και υπάρχει μια κατάσταση όπου οι χώρες περνάνε σε μια νέα ε, πραγματικότητα. Εμείς θα πρέπει να τις βοηθήσουμε να σταθεροποιηθούν, να δείξουμε την εμπειρία μας, την εμπειρογνωματοσύνη, διότι αυτοί δεν έχουν εμπειρία όσον αφορά αυτό που λέμε background, όσον αφορά το, το δημοκρατικό πλαίσιο. Σε αυτά εδώ λοιπόν τα πλαίσια υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να πούμε. Ήδη ελέγχθησαν εξάλλου ότι το θέμα του δημοκρατισμού θα πρέπει να σχετιστεί με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να έχει μια σημαντική θέση. Δεύτερη πτυχή όπως είπε η κυρία Ντεγκέζερ, ότι θα πρέπει να το σχετίσουμε το όλο θέμα σε σχέση με την ανάπτυξη. Μια προϋπόθεση. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Σημαντικό αυτό για να δημιουργήσει κανείς ένα χώρο μέσα στον οποίο η δημοκρατία θα μπορέσει να αναπτυχθεί. Αγώνας κατά της φτώχειας. Για το θέμα της υγείας, αγώνας για την υγεία, για την εκπαίδευση, όλα αυτά είναι πτυχέ που έχουν να κάνουν με ένα καλύτερο πεδίο ανάπτυξης δημοκρατία. Η οικονομική διακυβέρνηση, όλα αυτά στα πλαίσια μιας εξωτερικής πολιτικής πρέπει να συνδυαστούν. Όπως και η φτώχεια. Επίση να πω ότι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον ε, προπολογισμού που παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην κοινωνική των πολιτών ε, και οι κυβερνήσει των χωρών που είναι αυτές μέσα των οποίων μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να αναπτυχθεί η δημοκρατία. Επίσης να προσθέσω ότι κλείνοντας όπως έχουμε μια υπηρεσία για τις εξωτερικές υποθέσεις, υπάρχει μια υπηρεσία για τις τους υπηρεσίες των ανθρώπων και θα χρειαστεί οπωσδήποτε θα χρειαστεί ένας χώρος στον οποίο να υπάρχει κάποιος υπεύθυνο εκπρόσωπάς μας ο οποίος θα είναι συντονιστής για θέματα που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ θα καταθέσω μετροπολογία σε αυτό το πνεύμα στην έκθεση του κ. Σφένσον, η οποία πραγματικά πρέπει να την υποστηριχθεί από εμά. Και όπως πρέπει να την υποστηρίξουμε, οπωσδήποτε πρέπει να την εμπλουτίσουμε. Ευχαριστώ. Και εγώ θα πάρω το λόγο, λέει η Πρόεδρος. Τη στιγμή που έχουμε εδώ τον κύριο Σφένσον και τον κύριο Γκέρερο και τα άλλα μέλη της Επιτροπής που μου μιλήσανε σήμερα. έχουν υπάρχουν άτομα τα οποία φύγανε από τις χώρες όπου έγινε Επανάσταση, την Ισία, Λιβύη, έχουν πάει στην Λαπεντούσα, Φερρυπίνε, και προσπαθούν να μπουν στην Ευρώπη. Και οι χώρες ε, αρνούνται να εφαρμόσουν την οδηγία για άμεση υποστήριξη. Τι σκέφτεστε συνάδελφοι μήπως είναι επίγον το θέμα κάθε χώρα να δεχθεί κάποιους ανθρώπος, να είναι η δική μας συμβουλή για την οικοδόμηση της δημοκρατίας, δηλαδή να κάνουμε μια ποσόστοση κάθε χώρα. Να κάνουμε δηλαδή μια συμφωνία με αυτούς για κάποια χρόνια, ούτως ώστε να σταθεροποιηθούν οι δημοκρατίες. Η Νορβηγία σίγουρα μπορούσε να το κάνει, η Σουηδία, η Ισπανία επίσης και είναι η στιγμή την οποία πρέπει να δράσουμε. Αν θέλει τώρα η Επιτροπή να πάρει το λόγο για αυτή την έκθεση, παρακαλώ. Κάποιος άλλος από τις... την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων, όχι. Λοιπόν, άρα θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Σβένσο. Ευχαριστώ για όλες τις πολύ σωστές απόψεις που ε- παρουσιάστηκαν εδώ, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να τις λάβω υπόψη, υπόψη συγγνώμη, απλώς να αναγνωρίσω, κυρία Πρόεδρε, ε, εξεπλάγην. Διότι ότι γράφοντας ε, για αυτήν την δημοκρατία θα μπορούσα να γράψω πολύ περισσότερα από ό,τι έγραψα σε αυτό το μικρό α4 χαρτάκι. Εγώ συμφωνώ με όσα για τον εκδημοκρατισμό, επίσης για τις κοινωνικές, τεχνικές πτυχές, αλλά επίσης να πω ότι σίγουρα η Ευρώπη μπορεί να ανοιχθεί απέναντι σε αυτούς που έχουν περάσει λαμπετούσα. Και εγώ λυπάμαι ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύονται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, οι αναφορές δηλαδή ότι απευθύνεται κανείς σε αυτό το θέμα. Μιλάει για αυτούς τους ανθρώπους σαν ένα βάρος. Συχνά αναφέρεται ε, η έκφραση παράνομοι ε, μετανάστες. Κοιτάξτε να δείτε, δεν, δεν προφεύγει κανείς με νόμιμο τρέπο, τρόπο για να γλιτώσει τη ζωή του. Δεν πρέπει να τους αποκαλούμε έτσι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και προτείνω στον κύριο Σβένσον να πάμε στη Σουηδία μαζί και στη Νορβηγία για να επιτύχουμε ποσοστώσεις ε, προσφύγων. 10. Αποστολή παρακολούθησης των εκλογών στο Νίγηρα. Έχουμε ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Σαντιάγκο Φίσας Αξέλα, ο, οποίος παρακολούθησε τη διενέργεια εκλογών στο Νίγηρα και του δίνω το λόγο αμέσως, ευθύς αμέσως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να εντάξουμε στο πλαίσιο αυτή την ε, αποστολή παρακολούθησης. Όπως ξέρετε, ο Νίγηρας είναι μια χώρα, μεγάλη χώρα, το διπλό της Γαλλίας με 15 εκατομμύρια κατοίκους, 98% των οποίων είναι μουσουλμάνοι, μουσουλμάνοι μετριοπαθείς κυρίως στο ε, νότο και στο βορρά βρίσκονται οι Τουαρέγ και ορισμένες αραβικές φίλες. Ε, αγαπούν ιδιαίτερα τη ε, δημοκρατία. Είναι ένας ειρηνικός λαός, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για, ότι για μία ζώνη, τη ζώνη Αγαδές, η οποία δεν βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του Νίγηρα, αλλά την ελέγχει η Αλκάιντα. Υπ' αυτή την έννοια αποφασίστηκε να αποσταλεί μία επιτροπή για να ε, παρατηρήσει, να παρακολουθήσει εκλογές σε δύο γύρους. Όπως γνωρίζετε, η Αλκίνη απήγαγαν δύο Γάλλους, τους οποίους και φώνευσαν στη συνέχεια. Η Λέδη Άστον αποφάσισε ότι θα έπρεπε να αποσταλεί αυτή η ομάδα παρατηρητών για να δούμε πώς αντιμετωπίζει αυτή η χώρα την τρομοκρατία και να δούμε πώς μπορεί να ε, αποχωρήσει, μάλλον να, περάσει από τη δικτατορία στη δημοκρατία αυτό το κράτος. Ο πρόεδρος Τανζά έχει εκλεγεί δημοκρατικά και το Σύνταγμα επιτρέπει ε, δύο θητείες, πέντε συν πέντε χρόνια. Ο πρόεδρος ε, Τανζά, όπως ξέρετε, οργάνωσε ένα πραξικό που αρνήθηκαν όλα τα κόμματα εκτός από το δικό του καθώς και το συνταγματικό δικαστήριο. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Σελού έκανε ένα στρατιωτικό πραξικόπημα, αλλά για να επαναφέρει τη δημοκρατία. Άρα έγιναν τοπικές εκλογές, ε, μεταρρυθμίστηκε το Σύνταγμα και διενεργήθηκαν και βουλευτικές εκλογές, καθώς και ο δεύτερος γύρος των προεδρικών. Αυτό μπορώ να πω είναι ότι αυτές οι εκλογές διενεργήθηκαν ε, μέσα σε συνθήκες ασφάλειας και ήταν απόλυτα διαφανής. Ίσως υπήρξαν ε, ορισμένα μικροπροβλήματα επιμελητιακού χαρακτήρα, αλλά υπήρξε διαφάνεια και αυτό μπορούμε να πούμε ότι ίσχυσε και στις βουλευτικές ε, καθώς και στις προεδρικές εκλογές. Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε ήδη παραστεί και μεταξύ 5 Ιανουαρίου και 5 Απριλίου επανήλθαν. Δεν απεστάλησαν παρατηρητές βραχυπρόθεσμα και εμείς δεν αποστήλαμε καμία αποστολή για λόγους ασφάλειας. Οι παρατηρητές μας συμμετείχαν σε όλες τις περιφέρειες εκτός από το Αγκαντές και διενεργήθηκαν με απόλυτη, υπό απόλυτη διαφάνεια οι εκλογές. Ο Σιφούμα Αμαντού εξελέγει με 58% έναντι του Σενή Ουμαρού που ήταν ο υποψήφιος του κόμματος που είχε υποστηρίξει τον πρόεδρο, ο οποίος είχε κάνει αυτό το πραξικόπημα. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η χώρα θέλει να εκδημοκρατιστεί και χρειάζεται αναπτυξιακή βοήθεια για να μπορέσει να ανταποκριθεί και να καταπολεμήσει τους Κίμι στο βορρά της χώρας. Αυτά τα φύλλα θέλουν να επιζήσουν και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δοθεί αναπτυξιακή βοήθεια. Μιλήσαμε για την Αίγυπτο, Λιβύη και την Τινησία, γιατί προέκυψαν πολύ ε, νεκροί, αλλά στην περίπτωση του Νίγηρα δυστυχώς τα ΜΜΕ δεν ασχολήθηκαν με τη χώρα αυτή. Υπάρχει και ε, ανησυχία, μεγάλη ανησυχία από τις αρχές του Νίγηρα, δηλαδή το πώς, ε, τι έκφαση θα έχει η επανάσταση της Λιβύης μετά από την εκφρόνηση του Καντάφη. Υπάρχει όμως μία αποσταθεροποίηση της χώρας και πιστεύουμε ότι ο Καντάφη ποτέ δεν είχε εμπιστοσύνη στον στρατό του, ο οποίος αποτελείται από μισθοφόρους, γι' αυτό έχει, αποτελείται από διάφορες φυλές, γι' αυτό έχει μισθοφόρους που απαρτίζονται που μισθοφόρους και κυρίως του ΑΡΕΓ. Άρα δεν θέλουμε να σομαλοποιηθεί η χώρα. Γίνεται λόγος για μία κατάσταση αστάθεια στη Λιβύη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία ασταθή κατάσταση όπως ισχύει στο Σαχέλ ή στη Σομαλία. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ενδεχόμενες ερωτήσεις. Η κυρία Ντεκάιζερ. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον Σαντιάκο Φίσα, τον συνάδελφο, και να πω ότι χαίρομαι διότι Το θέμα είχε συζητηθεί επί μακρόν και όλα είχαν αίσιο πέρας. Έχω μία ερώτηση, δεν ξέρω αν είσαστε σε θέση να απαντήσετε. Μιλήσαμε για την προηγούμενη έκθεση ως προς το σύνδεσμο, τη διασύνδεση πολιτικής δημοκρατίας και οικονομικής βοήθειας και εδώ μας επισύρεται προσοχή στο ότι αν δεν υποστηρίξουμε τη χώρα θα υπάρξει μία αποσταθεροποίηση. Να ο συσχετισμός πολιτικής και οικονομικής δομής. Ως προς τα κριτήρια αποδοχής ε, και την ε, αποστολή των παρατηρητών δεν έχουμε απεριόριστα κονδύλια Όταν ε, μιλούσαμε για το Νίγηρα εδώ και μερικούς μήνες και την παρουσία της Αλκάιντα ε, Θα ήθελα να ρωτήσω πώς ε, κρίνεται ότι πρέπει, μιλάμε για αποστολή, για μια αποστολή που θα πρέπει να προωθηθεί και από την άλλη πλευρά μιλάμε για μη αποσταλή, αποστολή, δηλαδή σαν να παλινοδούμε. Και μένα με ρωτήσαν κατά πόσο ε, θα ήμουν επικεφαλής αυτής της αποσταλής. Μετά μου είπαν ότι θα ακυρωθεί για λόγους ασφάλειας και μετά έλαβαν την απόφαση να αποσταλεί. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε την εκλογική διαδικασία υπό δυσίωνες συνθήκες. Εν πάση περιπτώσει, διενεργήθηκαν οι εκλογές υπό διαφανείς συνθήκες. Επίσης, όμως, υπάρχει ένα πολιτικό ε, μήνυμα που πρέπει να αποσταλεί υφίσταται η χώρα αυτή τη μάστιγα της τρομοκρατίας, ο οποίος δεν μπορεί να καταπολεμηθεί. Ακόμα και σε αυτή τη μεταβατική φάση προς τη δημοκρατία από τη δικτατορία έγινε παραδειγματικά, υποδειγματικά. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε το ότι ευχαρίστησαν ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό μας συγκίνησε ιδιαίτερα. Επίσης έγιναν ορισμένες δηλώσεις υποστήριξης σε ώρα υψηλής τηλεθέασης, στην τηλεόραση και πολύ με ευχαρίστησαν γιατί ήμουν παρόν και τους υποστήριξα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα που αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες και έχουν χάσει πολλές επενδύσεις, διότι πολλές επιχειρήσεις δεν θα επενδύσουν στον Ήγηρα γιατί φοβούνται. Δεν μπορούν να προστατεύσουν τους εργαζόμενους τους και πολλές μη κυβερνητικέ επανέρχονται στη βάση τους για αυτό το λόγο. Τι θα κάνουμε. για αυτή την ε, δύσκολη περιφέρεια. Στη περιφέρεια του Σαχέλ μπορούμε να συγκρίνουμε την κατάσταση με τη Σομαλία, το Πακιστάν ή το Αφγανιστάν. Όμως ο ντόπιο πληθυσμός δεν έχει ενταχθεί στις δομές της Αλκάιντα, δηλαδή ε, πουλάνε μία γίδα, τι κάνουν, δεν έχουν ενταχθεί, αλλά πουλάνε τη γίδα τους τρεις φορές ακριβότερη σε ένα μέλος της Αλκάιντα. Ενώ σε έναν λευκό ή σε οποιονδήποτε άλλο την πουλούν πολύ φτηνότερα. Είναι ε, ένα θέμα, πρόκειται για ένα θέμα μέσω μακροπρόθεσμο. Θα πρέπει να υπάρχει στρατιωτική κατάρτιση, να προωθηθούν εξοπλισμοί και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη συγκυρία αυτή, διότι αφορά και τη Μαυριτανία και το Τσαντόχι μόνο το Νίγηρα. Πρόκειται για ένα θέμα ύψης της σημασίας για την Ευρώπη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμμετείχα στην αποστολή στην Ουγγάντα σαν παρατηρητρία. Ε, με, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η έκθεση για τις ε, ε, εκλογές στον Ήγερα. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος εκεί ε, έχει αυτή την εμπειρία ότι το είδαμε και στο Μαλί ότι δεν, οι στρατιωτικοί δεν σέβονται συχνά τα αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτό που ήθελα να σας πω, μόλις σας άκουσα για την ανάπτυξη σε, αυτή, σε αυτό το μέρος της χώρας που, όπου υπάρχουν δυνάμεις κατοχής, θα ήθελα να πω ότι η παρουσία σε αυτή τη ζώνη των πολιεθνικών η Αρεβά για παράδειγμα, και άλλες, έχουν μεγάλη ευθύνη για αυτές για τις δραστηριότητες τους, ουράνιο, κάτω από απίθανες συνθήκες, φοβερά σκληρές για τον κόσμο, η αίσθηση που έχει ο κόσμος εκεί ότι τους ε, ξεπουπουλιάζουν, τους παίρνουν όλο τον πλούτο και οι κάτοικοι σε αυτή τη ζώνη κάνανε όπως λέτε κάποιο εμπόριο και κάπως ε, κάνανε δεκτή την εκεί παρουσία. Έχουμε όμως η δραστηριότητα αυτών των πολυεθνικών, οι επιπτώσεις της οι δραστηριότητες των οποίων όμως έχουν επιπτώσεις οι οποίες δεν αποβαίνουν υπέρ των κατοίκων. Ήθελα να επιμένω σε αυτό το θέμα. Μιλάμε για ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει να γίνει κατανόητη. Μιλάμε για ανάπτυξη, αλλά να μην ε, γδέρνουμε τους Αφρικανούς, να μην. Εγώ ε, Γαλλίδα, είμαι και ξέρω προς τι, ε, τι εξυπηρετεί αυτό το ουράνιο. Το ουράνιο αυτό βοηθάει την ε, ανεξαρτησία, της, ε, την ενεργειακή ανεξαρτησία της Γαλλίας εις βάρος αυτού του λαού. Ε, το έχω κατανοήσει. Ξε, απ' τη μια έχουμε τον κόσμο του Νίγηρα και από την άλλη του ΑΚΜΗ υπάρχει μια αντιπαράθεση. Αλλά ξέρετε, αντιδρά και ο κόσμος. Δεν ζητούν ντε και καλά να τους βοηθήσουμε, αλλά αυτό που ζητούν είναι να είναι ανεξάρτητοι, να μπορούν να διαχειριστούν οι ίδιοι τον τόπο τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ροντ έχει το λόγο. Από την υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων από την υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων για το τμήμα που έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις σε σχέση με αυτά που είπε ο εισηγητές για τις δυσκολίες που υπήρχαν. Υπήρχε ένα πρόβλημα ε, με την ε, ασφάλεια αλλά και τη θέληση να βοηθήσει κανείς την, τον Ήγερα για αυτή την δημοκρατική διαδικασία με κάποιους περιορισμούς που τα ανέφερε ο μιλτής. Απλώς να πω ο, ή, για κάποια δήλωση θα ήθελα να πω ότι για μας ήταν μια, ε, ένα πέρασμα επιτυχημένο ε, με αξιοπιστία μια δημοκρατική διαδικασία. Όλοι οι υποψήφοι αναγνώρισαν το, τον τρόπο της διαδικασίας ήταν ε, σωστός. Αυτό είναι σπάνιο. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό που και τις δυσκολίε που υπάρχουν και όλοι ξέρουν σε όλες τις χώρες γύρω από τον Ήρα κυρίως όσον αφορά την δημοκρατική διακυβέρνηση είναι σωστό να υπογραμμίσουμε ότι η διαδικασία εκδημοκρατισμού είναι πετυχημένη. Σκέφτομαι όμως και το Μπενίν και άλλες χώρες όπου, οργανώ... Ε, όπου δεν οργανώθηκαν εκλογές οι οποίες όμως δεν ήταν τόσο επιτυχημένες όσο στον Ήγερα. Ε, υπογραμμίζει κανείς συχνά, αναφέρονται συχνά τα κακό κείμενα και όχι τα καλός. Ε, Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Ναι, για να δώσω τρόπον την κάποιες απαντήσεις στους συναδέλφους. Να υπογραμμίσω τη θέληση του Πρόεδρου Σαλού να, οδη προχωρήσει σε εκδημοκρατισμό. Και μιλήσαμε για το πέρασμα στην Προεδρία του νέου Πρόεδρου. Και στο Μπενίν έγινε, είχαμε την ίδια διαδικασία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Θέσεων που ήταν παρόν του είπε μήπως θα πρέπει να γίνει μια αναβολή για μια μέρα γιατί υπήρχε θέμα συνταγματικό. Ε, και ήθελε γρήγορα, γρήγορα να φύγει ο, ο παλιός πρόεδρος, το οποίο δείχνει ότι περνάμε σε, μια πιο, σε ένα πιο δημοκρατικό κλίμα. Έχουμε να κάνουμε με φτωχέ χώρες είναι μια από τις στοχότερες στον κόσμο, αλλά απ' την άλλη σε πρώτες ύλε είναι από τι πιο πλούσιες. Έχει χρυσό, ουράνιο, αλλά και πετρέλαιο. Είναι λοιπόν σαφέστατο ότι για το σύνολο της επικράτης ότι έχει, ε, έχει τέτοιους πόρους που θα μπορούσαν ε, να θα μπορούσαν, είναι εκμεταλλεύσιμες και αυτό μπορεί να ελκύσει επενδυτές. Και αυτό είναι σημαντικό για την ανάπτυξη της χώρας αυτής. Η παρουσία τώρα των Κινέζων αλλά και άλλων χωρών Ξέρουμε ότι ο Νίγερας είναι σημαντικός χώρος. Ο ποταμός είναι πολύ σημαντικός και εκεί έγινε και μια καινούρια γέφυρα από τους Κινέζους. και φυσικά το κάνουν πιο γρήγορα από εμά. Ξέρετε, οι διαδικασίε και είναι πιο, απλές, πιο απλοποιημένε. Δεν υπάρχουν συστήματα δημοσίων προσφορών. και λέγεται ας πούμε ε, μας είπαν εκεί πέρα ότι προτιμούμε τους Κινέζους, οι Κινέζοι είναι απο, αποτελεσματικοί, γρήγοροι ενώ δεν γίνεται το ίδιο με τους ε, ε Ευρωπαίους. Ε, θα πρέπει όμως να πάρουμε μέτρα ούτως ώστε να αποφύγουμε αυτό το dumping λεγόμενο που αποβαίνει βάρος των Ευρωπαίων. Τη στιγμή μάλιστα που εμείς συμβάλλουμε και βοηθούμε με πολλά κονδύλια. Ευχαριστώ. Κλείνουμε και αύριο στις 9 στην ίδια αίθουσα με νέα προεδρία.